Η ημερήσια διάταξη σας ε, έχει κατατεθεί και το πρώτο σημείο της ε, ημερήσιας διάταξης είναι έγκριση της ε, ημερήσιας διάταξης. Έχετε επιφυλάξεις ή παρατηρήσεις όσον αφορά την ημερήσια διάταξη. Από ό,τι φαίνεται όχι. Τώρα, μια τεχνική επισήμανση. Βρισκόμαστε σε έναν νέο χώρο συνεδριάσεων. Αν λοιπόν ε, θέλετε να βάλετε τις ε, κάρτες σας ε, μέσα στην ΟΠΗ, θα φανεί και ο αριθμό τη κάρτα. Τώρα, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θα ήθελα να σα ανακοινώσω σε σχέση με το σημείο υπαριθμών 4 τη ημερήσια διάταξη ότι πρόκειται για την παρουσίαση τη ε, ειδική έκθεση ε, του ε, κυρίου Διαμαντούρου. Γνωρίζετε περί τίνο πρόκειται. Πρόκειται για την διακριτική μεταχείριση των διερμηνέων. των διερμηνέων θα θέλαμε λοιπόν να καλωσορίσουμε τον ε, κύριο Διαμαντούρο και θέλω να σας πω ότι είναι μεγάλη χαρά για μένα το ότι μπορώ να καλωσορίσω τον ε, κύριο Διαμαντούρο. Ο κύριος ε, Διαμαντούρος θα μας παρουσιάσει ορισμένα στοιχεία της ειδική του έκθεσης που αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες διερμηνείς του διερμηνείς ε, freelance. Ε, Κυρίως πρόκειται για την ε, πρόσληψή τους στην Κομισιόν. Θέλαμε να έχουμε μία σύντομη έκθεση για αυτό το θέμα. Δυστυχώς δεν εγκρίθηκε αυτή από τη διάσκεψη των Προέδρων πριν από μία εβδομάδα στο Στρασβούργο. Ως εκ τούτου το σημείο υπαριθμών 5 ε, που αφορά την παρουσίαση του κυρίου Μαρτίνες Μαρτίνες Καταπίτη, εκτός εάν ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες ε, θέλει να λάβει παρόλα αυτά το λόγο επί του θέματος που βεβαίως έχει αυτό το δικαίωμα ε, λόγω του ότι δεν εγκρίθηκε η έκθεση πρωτοβουλία, ως εκ τούτου καταπίπτει και το αίτημα για ε, παρουσίαση της υπόθεσης. Όσον αφορά τώρα τα σημεία 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 15, αύριο θα έρθουν ε, οι ε, αναφέροντες. Πρόκειται και για τα δηληστήρια στο Μπιλπάο. Εκεί επ' αυτού θα εμφανιστεί ο αρμόδιος υπουργός θα ήθελα να σας υπενθυμίσω στα 5, 35, 38 τα σημεία αυτά διαγράφηκαν από την ημερήσια διάταξη και η ψηφοφορία σχετικά με την τοποθέτηση της κυρίας Σίνακ και της κυρίας Άουγγελ. Αυτή η συνεδρία θα γίνει αύριο με αυτά ε, την συνεδρία των συντονιστών. Η συνεδρία των συντονιστών θα ξεκινήσει στις 9 και η ψηφοφορία στις 10. Θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παρακαλέσω να φέρετε αύριο και τις ε, κάρτες σας για την ψηφοφορία. Έχουμε μια ολόκληρη σειρά ψηφοφοριών που σημαίνει ότι θα πρέπει να φέρετε τις κάρτες σας μαζί σας. Κύριε και κύριοι, θα ήθελα να σας κάνω μία ακόμα ανακοίνωση. Ο Σερ Ρόμπερτ. Πρόεδρε, θα ήθελα να γραφτεί στα πρακτικά πριν να προχωρήσουμε και φαντάζομαι θα το γνωρίζετε αυτό γιατί έχω στείλει ένα email στη γραμματεία του ΕΛΚ ότι στην ψηφορία αύριο που κατά πάσα πιθανότητα ε, θα είναι το λιγότερο επίμαχη, ας το πούμε έτσι, θα υπάρξει διάσταση απόψεων και γι' αυτό θα ήθελα να εφαρμόσετε ε, πολύ προσεκτικά τον κανονισμό 179. Ξέρω ότι αναφέρθηκε αυτό στην ιδέα των συντονιστών και το στηρίζω επιφύλακτα. Άρα δηλαδή δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και έχουμε ήδη ενημερώσει 24 ώρες πριν από την ψηφοφορία. Πρόεδρος, ε, γνωρίζω πολύ καλά το θέμα και συμμερίζομαι βεβαίως ε, την ε, άποψή σας ότι το όντι ε, είναι δυνατόν να υπάρξει διάσταση απόψεων για το θέμα αυτό. Εμείς λοιπόν την όλη διαδικασία ε, θα την εφαρμόσουμε σύμφωνα με το άρθρο 178. Ο κύριος Μαρτίνες ε, Μαρτίνες θα ήθελα ως διαδικαστικό να προτείνω να μην δεχθούμε την άποψη της διάσκεψης των Προέδρων, η οποία διάσκεψη απέρριψε τη δυνατότητα να υπάρξει μια έκθεση εν είδη συνέχειας μετά από αυτήν που θα παρουσιάσει ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής. Αυτό είναι ένα πολύ απλό θέμα που θα μας παρουσιάσει ο Διαμεσολαβητής και ε, το Κοινοβούλιο έχει τοποθετηθεί επ' αυτού. Αυτό που θα πρέπει να κάνουμε στην Ολομέλεια είναι να στηρίξουμε το διαμεσολαβητή, δηλαδή ε, να στηρίξουμε έτσι κι αυτό που το Κοινοβούλιο έχει ήδη αποφασίσει, το οποίο όμως δεν δέχεται η Κομισιόν η απόφαση αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από την Κομισιόν. Άρα δηλαδή είναι πάρα πολύ απλό το θέμα. Το μόνο που απομένει είναι να απευθυνθούμε στην Κομισιόν και να τη πούμε ότι θα θέλαμε να ε, εφαρμόσει η Κομισιόν την απόφαση του διαμεσολαβητή ακριβώς όπως το κάνει το Κοινοβούλιο. Εξάλλου να πω ότι είναι μια ειδική περίπτωση και μην ξεχνάμε ότι ο σονούπο ε, επίκειται και η ε, πανεκλογή του διαμεσολαβητή. Άρα δηλαδή αυτό σημαίνει ότι η ε, πρόταση του διαμεσολαβητή θα παραμείνει χωρίς καμία συνέχεια για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω λοιπόν ότι η δική μας Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει τη διαδικασία, να έχουμε μια σύντομη, σύνοπτη έκθεση, αυτή η έκθεση να κατατεθεί στη συνεδρίαση στο Στρασβούργο και να απευθυνθούμε στην Επιτροπή ή αν θέλετε στη διάσκεψη των Πρόεδρων και εφόσον κρυθεί απαραίτητο και στο Προεδρείο για να συζητηθεί το θέμα. Γιατί το θέμα αυτό είναι ε, ιδιαίτερο. Είναι ειδική περίπτωση όπως λέει και η απόφαση. Η απόφαση λέει ότι δεν θα πρέπει να εισαχθούν περισσότερες ε, αποφάσεις εκτός βέβαια αν υπάρξουν ειδικέ περιπτώσεις. Με πάση περιπτώσει δεν θα έχουμε συζήτηση στο Κοινοβουλίο, θα είναι απλά μια ψηφοφορία. Νομίζω όμως ότι θα είναι πολύ σημαντική η ψηφοφορία αυτή και ως εκ τούτου απευθύνω έκκληση σε εσά κύριε Πρόεδρε να συζητήσουμε για το σημείο υπαριθμών 5 και να αποφασίσουμε ότι θα συνεχίσουμε έτσι ώστε η έκθεση να συμπεριληφθεί στην έκθεση της ε, Ολομέλειας. Κοιτάξτε, εγώ προτείνω να μην συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Ε, την άποψή σας και ίσως ε, θα πρέπει αύριο ε, στις συνεδρίες των συντονιστών να συζητήσουμε για το θέμα αυτό, για το τι είδους διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουμε για να επιδιώξουμε κάποια αποτελέσματα. Συμμερίζομαι λοιπόν την άποψή σας και επιτρέψτε μου να κάνω και μία άλλη ανακοίνωση. Η αναφορά 939 Εκεί οι αναφέροντες είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με ε, την απόφαση. Πρόκειται για την καταβολή συντάξεων στο Λουξεμβούργο. Ε, και αναφέρομαι στην 616 κάθετος 05 1173-03 και πρόκειται επίσης ε, και για την αναφορά 80 λέει ο πρόεδρος και υπάρχει και η πρόταση αυτή η αναφορά 80 κάθετος 06 αυτή να επανέλθει εκ νέου. Και η 1265 κάθετος 07. Όσον αφορά την ομάδα Β, γνωρίζετε ότι πρόκειται για αναφορές οι οποίες μετά από γραπτή ενημέρωση κομισιών πρέπει να εξεταστούν. Τα μέλη της Επιτροπής κατέθεσαν την πρόταση. Τα σημεία ε, 58 59 να μην συμπεριληφθούν. Μήπως ε, θέλετε κάποια σημεία, κάποια θέματα της ομάδας Β να μεταφερθούν στην ομάδα Α. Αν ισχύει αυτό μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τη γραμματεία. Κατά τα άλλα, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Θα ήθελα να πω ότι μετά από πρόσκληση των αναφερόντων ε, ε, από πέρυσι πήγα... Πήγα στο Gated και στο Newcastle. Πρόκειται για μια χωματερή. Ε, τρεις ε, ευρωβουλευτές ε, ήταν ενημερωμένοι. Επ' αυτού εμφανίστηκαν η κυρία Φιώνα Χάου και ο βοηθός του Μάρτιν Κάλαχαν. Και αυτοί συμμετείχαν σε μία συζήτηση. Οι αναφέροντες λοιπόν είχαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την κατάσταση και κυρίως λόγω του ότι η χωματερή αυτή βρίσκεται πολύ κοντά στα σπίτια τους. Οι τοπικές αρχές έδωσαν λεπτομερείς πληροφορίες για αυτήν την υπόθεση, για το πώς ε, ακριβώς ε, δημιουργήθηκε αυτή η χωματερή. Εγώ μάλιστα ε, δέχτηκα μία πρόσκληση από το Δημοτικό Συμβούλιο του Νιουκάσιλ και μετά από την πρόσκληση του Συμβουλίου που σας είπα μεταβήκαμε και επιτόπου γραπτή έκθεση προτιθέμεθα να σας καταθέσουμε σύντομα. Ο Σερ Ρόμπερτ έχει το λόγο. Πρόεδρε, δεν θέλω να αναφερθώ σε πάρα πολλέ λεπτομέρειε από αυτού, αλλά θα ήθελα να πω το εξή, ότι η αρχή σχετικά με αυτή την επίσκεψη στο Νιου Κάστιλ θα μου επιτρέψετε να την επαναλάβω. Σύμφωνα λοιπόν με τι διαβουλεύσει που είχαμε συντονιστές συντονιστέ άλλων ομάδων και με άλλα μέλη τη Επιτροπή, πρέπει να σα πω ότι δεν είχαμε ιδέα για αυτή την επίσκεψη. Ούτε και η Επιτροπή, αλλά ούτε και οι συντονιστέ εκλήθησαν να τοποθετηθούν. Ένα συνάδελφό μου από το Ηνωμένο Βασίλειο ήρθε και με βρήκε για να μάθει τι γινόταν, γιατί ούτε και κύριο ήξερε τίποτα και εγώ, ούτε και εγώ μπορούσα να του πω τίποτα γιατί και εγώ δεν ήξερα. Ω εκ τούτου, Πρόεδρε, κάτω από αυτέ τι συνθήκε δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Γι' αυτό λοιπόν, ε, για να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, θα ήθελα να επιμείνω πρώτον από τώρα μέχρι στο απόλυτο δίνεκε, εν σίγουρα μέχρι τι επόμενε εκλογέ, για τι επισκέψει θα πρέπει να υπάρχουν διαβουλεύσει με του συντονιστέ. Και ελπίζω και να υπάρχουν διαβουλεύσει με την αρμόδια επιτροπή πριν ληφθεί οποιαδήποτε τέτοια μορφή απόφαση. Ευχαριστώ για αυτά τα σχόλια. Νομίζω ότι εξηγήσαμε την τελευταία συνεδρίαση τι ακριβώς συνέβη. Υπάρχουν άλλα σημεία από τα διάφορα? Όχι. Ωραία. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Διαμαντόρες. Διαμαντούρο, συγγνώμη. Good morning. Chairman. Καλησπέρα σας όλοι. Καλησπέρα κύριε Σερ Ρόμπερτ. Πάντα αισθάνεται κάποιος λίγο ανησυχεί όταν έρχεται εδώ ενώπιον της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να κάνω μία σύντομη παρουσίαση των επιχειρημάτων μας. Ε, εμφανίζομαι μπροστά σας όταν υπάρχει ειδική έκθεση στο Κοινοβούλιο. Ε, η ειδική έκθεση είναι το απότατο όπλο του διαμεσολαβητή. Ο θεσμός του διαμεσολαβητή ε, στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο δεν ε, υπάρχει, αλλά δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει νομικά δεσμευτικές αποφάσεις. Χωρίς αυτή τη δυνατότητα, οι διαδικασίες του διαμεσολαβητή φυσικά είναι πιο ευέλικτες από των δικαστηρίων και τα κριτήρια είναι πολύ πιο ευρύ, ευραία. Επομένως, οι πολίτες έχουν μια πραγματική επιλογή μεταξύ μιας δίκης, μιας δικαστικής δηλαδή διαδικασίας και μιας μη δικαστικής διαδικασίας και κάθε διαδικασία έχει τις, ε, τα θετικά της και τα αρνητικά της. Εμείς βασιζόμαστε στην πυθό, στην ικανότητα να πείσουμε μέσω επιχειρημάτων, βάσιμων επιχειρημάτων, μερικές φορές μέσω της διαφήμισης και μέσω της, ε, της γνώμης του κοινού. Μέσα στα 16 τελευταία χρόνια ε, η στάση του διαμεσολαβητή δείχνει την δυνατότητα συνεργασίας που έχουμε. Ε, ένα τμήμα της εξουσίας του είναι αυτή η ειδική έκθεση που κάνει στο Κοινοβούλιο. Το επόμενο βήμα που μπορεί να είναι αυτή η ειδική έκθεση για μια αναφορά ε, συχνά εξαναγκάζει τον ενδιαφερόμενο, το θεσμικό όργανο να αλλάξει την αποφασή του. Ε, οι ειδικέ εκθέσεις δεν παρουσιάζονται πολύ συχνά, μόνο για πολύ σημαντικά θέματα, ε, επί των οποίων το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να βοηθήσει το ε, εν λόγω θεσμικό όργανο να αλλάξει την αποφασή του. Ως πολιτικό όργανο το Κοινοβούλιο είναι κυρίαρχο για να αντιμετωπίσει όπως θέλει τις ειδικέ εκθέσεις του διαμεσολαβητή. Ελπίζω όμως ότι σε ό,τι αφορά μια ειδική έκθεση, το Κοινοβούλιο πάντα λαμβάνει υπόψη το δικαίωμα να στραφεί προς το διαμεσολαβητή και αυτό είναι σημαντικό στοιχείο, ε, σημαντικό όπλο αν θέλετε της ηθαγενειάς μας. Ας ε, στραφώ τώρα στην ειδική έκθεση που παρουσιάσα στο Κοινοβούλιο στις 4 Δεκεμβρίου του 2008. Ο αναφέροντας δούλεψε για τα κοινοτικά όργανα παραπάνω από 35 χρόνια ως freelance διερμηνέας. Στην ιδιόγνωση που χρησιμοποιούμε για τους ε, διερμηνείς ήταν ε, διερμηνέας freelance ACI. Κάποια στιγμή αποφασίστηκε τα όργανα να, μην προσλαμβάνουν πια τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών. Γιατί, Γιατί ε, οι υπόλοιποι υπάλληλοι της κοινότητας δουλεύουν μέχρι τα 65 και επομένως ε, και οι freelance διερμηνείς καλύπτονται από αυτές τις διατάξεις. Εν συνεχεία, κάποιοι ε, freelance διερμηνείς ε, προσέφηγαν στο πρώτο δικείο το 2004. Το 2004 το πρωτοδικείο αποφάσισε ότι η Κομισιόν είχε άδικο να θεωρήσει ότι το όριο σταξιοδότησης για τους freelance διερμηνείς ήταν το ίδιο με των υπολείπων υπαλλήλων της κοινότητας. Δεν είναι το σωστό επιχείρημα αυτό, ε, η σωστή βάση για να κρίνουμε έναν freelance ε, διερμηνέα. Με βάση τον αναφέροντα, ο οποίος ήταν έναν των 65, η Κομισιόν ε, δεν συμμορφώθηκε και μετά την απόφαση του πρωτοδικίου να τον προσλάβει. Γι' αυτό ακριβώς στάθηκε προς εμένα και υπέβαλε μία αναφορά. Η Κομισιόν είπε για αυτή την αναφορά ότι μετά την απόφαση του πρώτοδικίου, επανέφερε την πολιτική που είχε πριν από το 1999. Επίσης είπε ότι θα συνεχίσει να συμμορφώνεται με αυτή την πολιτική περιμένοντας την απόφαση του ΔΕΚ, γιατί η Κομισιόν έχει προσφύγει στο ΔΕΚ, που με σκοπό να ανατραπεί η απόφαση του πρωτοδικίου. Όμως μετά μια ε, προσεκτική ανάλυση της πολιτικής της Κομισιόν, ε, με οδηγήσει να, καταλήγω, να καταλήξω ότι δεν συμμορφώνεται με την απόφαση του πρωτοδικίου. Η Κομισιόν δήλωσε ότι είχε δικαίωμα να προσλάβει freelance διερμηνείς με βάση, όπως λέει, τις ανάγκες της υπηρεσίας, λαμβάνοντας υπόψη τον γλωσσικό συνδυασμό, την διαμονή και γενικά τις επιδόσεις, τις ικανότητες του διερμηνέα. Είπε ότι έχει το δικαίωμα να αντιμετωπίσει διαφορετικά τους διερμηνείς αν των 65, γιατί με βάση τις ανάγκες υπηρεσίας είναι υποχρεωμένη να δώσει ευκαιρίες σε νέους ε, διερμηνείς. Η Κομισιόν τόνισε σε αυτό το πλαίσιο ότι τα θεσμικά όργανα υποστηρίζουν διαμακρών την εκπαίδευση των νέων ε, συναδέλφων, ε, τους δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουν αρκετή πείρα και με αυτόν τον τρόπο να αυξήσουν τη δυνατότητα να προσθέσουν νέες γλώσσες στο γλωσσικό του ε, συνδυασμό. Σε σχέση με την από αυτά που λέει η Κομισιόν, θα ήθελα να πω ότι η αρχή του άρθρου 21 ε, της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων για μη ε, διάκριση λόγω ηλικίας είναι βασικό στοιχείο του κοινοτικού δικαίου. Δηλαδή τα άτομα δεν θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε διαφορετικά λόγω της ηλικίας εκτός και αν αυτή η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται ε, όπως δει. Η Κομισιόν όμως πιστεύω ότι ανοιχτά παραδέχτηκε ότι μεταχειρίζεται διαφορετικά τους διερμηνείς ανά των 65. Θεωρώ λοιπόν ότι η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να μας δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι αυτή η διαφορετική μεταχείριση δικαιολογείται. Ότι συντρέχουν λόγοι για αυτήν. Δέχομαι ότι το συμφέρον που αναφέρει η Κομισιόν, δηλαδή η εκπαίδευση μιας νέας γενιάς διερμηνέων, είναι ένα πραγματικά θεμητό συμφέρον. Παρ' όλα αυτά αναφέρω ότι η Κομισιόν δεν μας έδωσε επαρκή στοιχεία για να αποδείξει ότι όντως έπρεπε να σταματήσει να προσλαμβάνει τους διερμηνείς, freelance διερμηνείς άνω των 65 για να προστατεύσει αυτό το θεμητό και νόμιμο συμφέρον. Επιπλέον η Κομισιόν δεν απέδειξε ότι υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στα ε, δικαιώματα των διερμηνέων άνω των 65 και τα δικά της θεμητά συμφέροντα. Επίσης ε, σημειώνω ότι μια πολιτική για την δημιουργία μιας νέας γενιάς διερμηνέων θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να εξασφαλιστεί και με λιγότερο επαχθή μέσα που να βαραίνουν όχι μόνο δηλαδή τους διερμηνείς ανά των 65. Γι' αυτό πιστεύω ότι η Κομισιόν δεν δικαιολόγησε επαρκώς ε, τη μεταχείριση. Προτείνω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να εγκαταλείψει την πολιτική διακριτικής μεταχείρισης ε, ε, των διερμηνέων ανά των 65 και να ε, προσφέρει ε, εύλογη ε, αποζημίωση προς τον αναφέροντα λόγω του ότι το μεταχειρίστηκε διαφορετικά. Πρόκειται για μια φιλική λύση. Η απάντηση της Κομισιόν είναι ότι το ΒΕΚ πρόσφατα ακύρωσε την απόφαση του πρωτοδικίου. Η Κομισιόν είπε ότι η αρχική ερμηνεία των κανόνων, όπου δεν προσέφερε καθόλου δουλειά στους άνω των 65, ήταν σωστή και ότι θα εξακολουθήσει να είναι σωστή μέχρι μια απόφαση ε, από ένα ευρωπαϊκό δικαστήριο, από το ΔΕΚ δηλαδή, να προκύψει που να ανατρέψει αυτά τα στοιχεία. Είναι επομένως υποχρεωμένη να εφαρμόσει μια πολιτική μη πρόσληψης ανθρώπων που έχουν ε, συμβόλια και φτάνουν ε, την ηλικία των 65. Αγαπητοί συνάδελφοι, εξέτασα με προσοχή την απόφαση του δικαστηρίου, του ΔΕΚ. Το, ΔΕΚ ακύρωσε την απόφαση του πρωτοδικίου γιατί το πρωτοδικείο θα έπρεπε κανονικά να μην θεωρήσει παραδεκτή την υπόθεση αυτή. Το ΔΕΚ δεν ε, αποφάνθηκε επί της ουσίας της υπόθεσης και επομένως δεν ε, είπε τίποτα για την νομική ερμηνεία της απόφασης του πρωτοδικίου. Η Κομισιόν σωστά είπε ότι πλέον δεν, είναι νομικά, δεν δεσμεύεται νομικά από την ακυρωμένη απόφαση του πρωτοδικίου. Παρ' όλα αυτά δεν εξήγησε γιατί δεν θα έπρεπε να επιλέξει να φτάσει με τα ίδια στα ίδια συμπεράσματα με αυτά στα, οποία, στα οποία έφτασε το πρωτοδικείο επί της ουσίας της υπόθεσης. Δεν συμφωνώ με το επιχείρημα ότι για νομικούς λόγους η Κομισιόν δεν έχει επιλογή παρά να σταματήσει να προσλαμβάνει τους freelance διερμηνείς άνω των 65. Πιστεύω, μάλιστα, ότι η Κομισιόν δεν προσλαμβάνει τους ε, διερμηνείς άνω των 65 γιατί επιλέγει να μην τους προσλάβει. Όπως ε, σημείωσα είπα, επίσης, το συμφέρον που επικαλείται η Κομισιόν στην νομοδότηση της, ότι πρέπει δηλαδή να δημιουργήσει ε, δυνατότητες για νέους διερμηνείς και να τους εκπαιδεύσει, είναι θεμητό συμφέρον. Παρ' όλα αυτά δεν είμαι πεπισμένο ότι μια πλήρης απαγόρευση της πρόσληψης των διερμηνέων άνω των 65 είναι αναγκαία για να πετύχει αυτό το θεμητό συμφέρον, αυτό το θεμητό σκοπό. Γι' αυτό θεωρώ ότι η Κομισιόν δεν κατάφερε να δικαιολογήσει την απαγόρευση πρόσληψης ε, των διερμηνέων άνω των 65. Αυτό αποτελεί ε, στοιχείο κακοδιαχείρισης. Τονίζω ξανά ότι τα πορίσματά μου για αυτή την υπόθεση είναι συμβατά με τις αποφάσεις και των δύο δικαστηριών του Πρωτοδικείου και του ΔΕΚ. Η ακύρωση της απόφασης του Πρωτοδικείου από το ΔΕΚ γιατί, γιατί η απόφαση αυτή αρχικά θα έπρεπε να θεωρηθεί παραδεχτή, μη παραδεχτή από το Πρωτοδικείο δεν σημαίνει ότι η ουσία των επιχειρημάτων του πρωτοδικείου δεν ισχύει. Το πρωτοδικείο αποφάσισε επί της ουσίας της υπόθεσης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι σε μια αντίστοιχη έρευνα, στην οποία αναφέρθηκε ο κ. Μαρτίνες Μαρτίνες, που έκανα για τις πρακτικές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την πρόσληψη των ε, freelance διερμηνέων άνω των 65, έκανα ένα σχέδιο σύστασης προς το Κοινοβούλιο και το αποτέλεσμα ποιο ήταν. Το Κοινοβούλιο δέχτηκε τη θέση μου, άλλαξε τι πρακτικέ του ό,τι αφορά την πρόσληψη των freelance διερμηνέων άνω των 65. Με αυτή τη θέση του, το Κοινοβούλιο ερμήνευσε του εφαρμοστέου κανόνε που είναι οι ίδιοι κανόνε, με διαφορετικό τρόπο, με τους, και είναι για, μιλάμε για κανόνε που θα έπρεπε να εφαρμόζει και η ίδια η Κομισιόν. Του εφάρμοσε όμω με τέτοιο τρόπο που δεν οδηγούν σε απαγόρευση τη πρόσληψη των διερμηνέων άνω των 65. Με αυτόν τον τρόπο ε, το Κοινοβούλιο ε, δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι έχει προβεί σε κακοδιαχείριση. Θα ήθελα να κάνω κάθε προσπάθεια για να βοηθήσω την ε, Κομισιόν να αποφύγει αυτή την κακοδιαχείριση, αλλά δεν νομίζω ότι αντέδρασε με θετικό τρόπο. Θεωρώ ότι αυτή η περίπτωση κακοδιαχείρισης που βασίζεται στη διάκριση λόγω ηλικίας αρκεί για να δικαιολογήσει την ειδική έκθεση που υποβάλλω στο Κοινοβούλιο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής και βεβαίως ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Είμαι στην διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινήσεις. <clears throat> Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την πολύ λεπτομεριακή παρουσίαση. Εξ ονόματος της Επιτροπής θα μιλήσει ο Τζόρτζι Δικάρ. Παρακαλώ. Euh, merci, euh, euh, πολύ, κύριε Πρόεδρε, άκουσα με μεγάλη προσοχή τις εξηγήσει που δόθηκαν από τον διαμεσολαβητή. Ε, πραγματικά εκφράστηκε πολύ καλά, εξέφρασε πολύ καλά ε, και περίεργασε πολύ καλά όλες τις ανταλλαγές που είχαμε με αυτόν. Θα ήθελα να υπενθυμίσω την κατάσταση έτσι όπως τη βλέπει η Επιτροπή από το 2000 μετά από την υπογραφή της σύμβασης με τους διερμηνείς freelance, ε, οι διερμηνείς συγγνώμη freelance έγιναν ACI. Και ε, σε συνέχεια άλλαξε το καταστατικό και εντάχθηκαν ε, στο, στο σύστημα που προβλέπει ο κανονισμός και το οποίο σημαίνει ότι μπορούν να επωφεληθούν από το κοινοτικό δίκαιο. Και από εκείνη τη στιγμή υπήρξε μια κίνηση ούτως ώστε να υπάρξει μια ευθυγράμμιση όσον αφορά τη μεταχείριση των παλιών freelance με αυτή των υπαλλήλων. Και εφόσον ε, συμπεριλήφθησαν σε αυτό το ε, σύστημα ίσης μεταχείρισης, οι προϋποθέσεις που ορίζονται στον κανονισμό εφαρμόζονται στους πρώην ε, διερμηνείς freelance. Και αυτό δεν ισχύει μόνο από νομική πλευρά αλλά και από πολιτική πλευρά. Δηλαδή από το 2000 έγινε μια τροποποίηση της σύμβασης και υπογράφηκε μια, η τροποποιημένη σύμβαση στα τέλη του προηγούμενου έτους που τέθηκε σε ισχύ το μήνα Σεπτέμβριο, δηλαδή πριν από λίγο μόνο καιρό και σε αυτή τη σύμβαση ε, στο μέτρο του δυνατού, γιατί η κατάσταση των διερμένων freelance διαφέρει αυτή των υπαλλήλων, αλλά ε, προσπαθήσαμε να ευθυγραμμίσουμε τις, εξομοιώσουμε τις συνθήκες εργασίας τους. Για παράδειγμα, οι υποτροφίες ε, κατάρτισης, οι οποίες προορίζονταν μόνο για τους υπαλλήλους, τώρα από, από αυτές μπορούν να αποφεληθούν και οι διερμηνείς freelance. Και το κάναμε επειδή θεωρήσαμε ότι από το 2000 ε, ε, το καθεστώς των freelance ε, εξομοιώθηκε με αυτό ή προσεγγίζει αυτό των υπαλλήλων. Και πιστέψαμε ότι εφόσον η σύμβαση αυτή ήταν σιωπηλή, τελικά θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Αυτή η ερμηνεία που δόθηκε ε, είχε δέχτηκε κάποιες ε, αντιδράσεις από ορισμένε χώρες και Ε, έγιναν κάποιες ε, θέσεις και επί της ουσίας αλλά και τυπικές. Ε, και εμείς ε, τελικά ενισχυθήκαμε στην άποψή μας ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί αυτή η σύμβαση. πιστεύω ότι κάναμε μια προσπάθεια πειθούς και θα αποφύγουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ε, νομίζω ότι φέραμε, κομίσαμε κάποια σημαντικά νομικά επιχειρήματα για να θεωρούμε ότι βρισκόμαστε θέλουμε δικαίω. Και ε, βεβαίως εάν ε, υπάρξει συνέχεια θα εξετάσουμε τη νέα κατάσταση. Tak, więc proszę Państwa, κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες, ο κύριος Μαυρομάτης, ο κύριος Ρόμπερτ Άτκινς. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ε, παρεμβάσεις. Και αν δεν υπάρχουν άλλες θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Ο κύριος Μαρτίνες Μαρτίνες. Thank uh, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω στους ε, συναδέλφους το εξής. Εγώ δεν ομιλώ μόνο ως μέλος της Επιτροπής, αλλά και με την ιδιότητά μου του Αντιπροέδρου του Κοινοβουλίου, αρμόδιου για την πολυγλωσία, δηλαδή αρμόδιος για οτιδήποτε έχει ε, σχέση με, τις, ε, με τη μετάφραση και τη διερμηνία στο Κοινοβουλίο και όλα αυτά τα λαμβάνω πάρα πολύ σοβαρά. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να μακρηγορεί κανείς ε, στο θέμα αυτό. Αυτό που έχουμε μπροστά μας είναι μία απόφαση, μία πράξη του διαμεσολαβητή που περιλαμβάνει σύσταση και για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν με απότερο στόχο να επιληθεί το θέμα που αφορά και στους ε, δύο οργανισμούς ή, για να το πούμε αλλιώς, είτε είναι δικαιολογημένο είτε όχι, και η δύο ή ο ένας εξ αυτών έχει αποφασίσει να μην προσφέρει εργασία στους ε, συναδέλφους διερμηνείς, του διερμηνείς για πάρα πολλά χρόνια. Η ε, στάση όμως του Κοινοβουλίου είναι τελείως διαφορετική από αυτήν την Κομισιόν. Δηλαδή το Κοινοβούλιο δέχεται τις προτάσεις ε, του διαμεσολαβητή και η Κομισιόν διαφωνεί. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα για αυτά που είπε στο τέλος ο εκπρόσωπος της Κομισιόν είπε δηλαδή ότι ελπίζει ότι θα προσφερθεί η δυνατότητα να επανεξεταστεί το θέμα και το καθεξής. Αλλά εγώ νομίζω ότι η πρώτη αντίδραση της Κομισιόν είναι ενδεικτική της έπαρσης που χαρακτηρίζει την Κομισιόν σε καθημερινό επίπεδο και σε όλα τα επίπεδα, σε καθημερινή βάση και σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή η Κομισιόν δεν δέχεται να πει ή να παραδειχθεί ότι κάτι που κάνει είναι λάθος. Η Επιτροπή αυτή, αυτή την ε, συμπεριφορά τη βιώνει καθημερινά, αλλά όχι μόνο η δική μας Επιτροπή και άλλες Επιτροπές νιώθουν το ίδιο. Η Κομισιόν δηλαδή πιστεύει ότι είναι υπεράνω του Θεού, υπεράνω όλων, υπεράνω πάντων. Δεν ισχύει όμως αυτό. Οι κανονισμοί το η εφταξία ισχύει και για το Κοινοβούλιο και για την Κομισιόν. Το Κοινοβούλιο εξάλλου είναι το κυρίαρχο όργανο της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και εμείς δεχτήκαμε αυτή την απόφαση. Θεωρούμε ότι έχουμε το καθήκον να στηρίξουμε το διαμεσολαβητή ως ε, ε, θεσμό που λαμβάνει κατά κανόνα τις αποφάσεις του με σωστό τρόπο. Πάντως εκείνο που έχει σημασία είναι να κατανοήσει κανείς ε, τις αποφάσεις του διαμεσολαβητή και να τις σέβεται. Αυτό βέβαια ισχύει για, την, ε, για το Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν ε, θεωρεί το Κοινοβούλιο είναι ένας κάποιος οργανισμός, κάπου βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ισχύει που δεν είναι στην, ε, στον παντοδύναμο αυτό οργανισμό που είναι η Κομισιόν. Ε, οι μουσουλμάνοι όταν αρχίζουν ε, να προσεύχονται στον Θεό τους, τον ε, αποκαλούν παντοδύναμε, πανταχού παρόντα. Μερικές φορές λοιπόν έχει κανείς την αίσθηση ότι <clears throat> και για όλους τους άλλους όταν προσφανούν την Κομισιόν θα πρέπει να ισχύει το ίδιο. Αυτό όμως δεν ισχύει. Σε αυτή την περίπτωση ισχύει το εξής ισχύουν τρία πράγματα. Πρώτον, είναι καθήκον μας να στηρίξουμε ε, τον διαμεσολαβητή, να δεχθούμε την απόφασή του. Δεύτερον, να συμπεριφερθούμε με τρόπο συνεπή με τη συμπεριφορά μας, με τις ε, αξίες μας. Και τρίτον, να δείξουμε στην Κομισιόν ότι και εκείνη οφείλει να συμβιβάζεται, να σέβεται θεσμούς όπως είναι ο διαμεσολαβητής που έχουν αρμοδιότητες για μας, για την Κομισιόν, για το Συμβούλιο, οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Ως εκ τούτου λοιπόν τις συστάσεις του διαμεσολαβητή τις ερμηνεύω ως σημαντικές, ουσιαστικές, επίγουσες και επουδενή δεν θα πρέπει να κόλληση εργούμε, να συμβάλλουμε και εμείς σε μια καθυστέρηση που δεν έχει καμία σχέση με, τις, με τη συνέπεια και με τις αρχές ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριος ε, Μαυρομάτης έχει το λόγο. Παρακαλώ. Τον ε, κύριο Διαμαντούρο, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, διότι όπως πάντοτε έχει αποδείξει ότι είναι πολύ συνεπής πρώτον στην παρουσία του στη δική μας την Επιτροπή και δεύτερον με την εργασία η οποία έχει πάντοτε ένα θέμα για συζήτηση τόσο πολύ ευρύ ώστε να μας ενδιαφέρει πάντα και όχι μόνο την Επιτροπή μας αλλά και τα 500 εκατομμύρια των ε, πολιτών που μας παρακολουθούν. Θα ήθελα ε, όπως και ο συνάδελφος ε, Μιγέλ είπε στο θέμα της πολυγλωσσίας ήμουν ο εισηγητής της πρώτης έκτασης για την πολυγλωσσία συνεργαστήκαμε άμεσα και με τον διαμεσολαβητή όπως και ήμουν και ο εισηγητής για τον διαμεσολαβητή. Εκτιμώ ότι όλες οι αποφάσεις οι οποίες έχουν ε, πάρθει εδώ και ήμουν από τους πρώτους που στήριξε το θέμα των διερμηνέων όταν ακόμα το 2005 υπήρξε κίνδυνος απολύσεων και απομακρύνσεων διερμηνέων και μείωσης των διερμηνέων για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξαιτίας δυσπραγίας οικονομικής. Ευτυχώς συγκρατήσαμε το θέμα αυτό και δεν υπήρξαν ούτε απομακρύνσεις αλλά απέναντίας Χρησιμοποιήθηκαν και νέοι διερμηνείς εκτός από τους freelance αλλά και ως μόνιμοι. Εκείνο που εκτιμώ είναι ότι κακώς βιαστήκαμε να πάρουμε μία απόφαση αν δεν έχει υπαρθεί ακόμα και ερχόμαστε σε αντίθεση βεβαίως με την Κομισιόν όσον αφορά αυτήν την σύσταση του διαμεσολαβητή που στηρίζει ο, ο συνάδελφος Μαρτίνες εδώ που θα ήθελα και εγώ προτού αυτή η θητεία να φτάσουμε σε ένα θετικό αποτέλεσμα για να δούμε τα προβλήματα που υπάρχουν, να λύσουμε ενδεχομένως, να υποβοηθήσουμε επίσης την Κομισιόν ώστε θέματα εργασιακού περιεχομένου και εργασιακά κυρίως που κατ' επανάληψη έχουμε συζητήσει αυτά τα πέντε χρόνια να έχουμε την δυνατότητα να τα στηρίξουμε μέχρι τέλους και πριν ακόμα από τις εκλογές. Φρονώ λοιπόν ότι η θέση του συναδέλφου του Μαρτίνες είναι θετική από προσωπικά εγώ θα την στηρίξω και εφόσον μπορούμε και εμείς ως Επιτροπή να κάνουμε στην πλειοψηφία το ίδιο θα ήθελα κύριε Πρόεδρε να έχουμε την δυνατότητα μιας νέας θέσης απέναντι στην Κομισιόν και η Κομισιόν να επανεξετάσει μαζί με τον διαμεσολαβητή το όλο θέμα μια και σήμερα τουλάχιστον υπήρξε μια ε, αν θέλετε από πλευράς ε, Κομισιόν διαφορετική θέση ή άποψη, αν δεν κάνω λάθο από την αρχική θέση την οποία είχε μέχρι τώρα και έτσι η οποία μας μεταφέρθηκε. Θα ήθελα λοιπόν και πάλι να στηρίξω το θέμα αυτό. Στηρίζω ανεπιφύλακτα την εργασία των διερμηνέων, είτε freelance είτε όχι. Είναι για μας θέμα πολυγλωσία που πρέπει να διατηρήσουμε κύριε Πρόεδρε με κάθε θυσία και κάθε τρόπο ώστε με την διεύρυνση που ενδεχομένως έρχεται να μην μας λείψει αυτό το πολύτιμο εργαλείο που για όλους πολύ σημαντικό σε αυτό το κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ο διαμεσολαβητής πάντα παρουσιάζει τα επιχειρήματά του με νυφαλιότητα και σαφήνεια και βοηθάει ανθρώπους όπως εγώ που δυσκολεύονται με, τις, με τους νομικούς δεδάλους. Κάποιες ερωτήσεις. Αν καταλαβαίνω την ουσία, η ουσία έχει και κάποια τεχνικά θέματα. Ή μάλλον ε, η ουσία περιλαμβάνει την απόρριψη για, λόγο, για λόγους τεχνικούς. Δεν κατάλαβα αν πιστεύει ότι είναι ουσιαστικό αυτό το στοιχείο ή δευτερεύουν στην αναφορά. Εγώ πλησιάζω τα 65 και όσο πλησιάζω αυτήν την ηλικία αντιστέκομαι όλο και περισσότερο σε αυτούς που θέλουν να μας ξεφορτωθούν εμάς τους πιο ηλικιωμένους. Πιστεύω ότι έχω όλες μου τις δυνάμεις και επομένως διερωτώ με. Α, δεν περίμενα να γελάσετε σε αυτό το σχόλιο που κάνω τώρα. Διερωτώ με. Αυτό το όριο των 65 αφορά όλους τους διερμηνείς όλους τους υπαλλήλους ή μόνο τους freelance, τους ACI. Και γιατί. Γιατί οι ACI θα μπορούσαν κάποια στιγμή, ας πούμε, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και μετά τα 65. Ποιος είναι, ο, λοιπόν, ποιο είναι το σκεπτικό της Κομισιόν και δεν τους προσλαμβάνει. Τρίτον, η κακοδιαχείριση. Είναι το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγεται. Η Κακοδιαχείριση προκύπτει από την απόφαση της Κομισιόν ή ότι το γεγονός ότι αγνοούν την σοφή σας απόφαση και αυτό ε, οδηγεί σε κακοδιαχείριση. Τέλος, οι συντονιστές της Επιτροπής αποφάσισαν πρόσφατα ότι δεν θέλουμε άλλες εκθέσεις από τώρα μέχρι τις ε, εκλογές. Το ερώτημα που προέκυψε μια και περιμέναμε τη δική σας έκθεση ήταν πόσο επίγον είναι αυτό το θέμα. Αν είναι επίγον, όντως θα πρέπει να το διεκπαιρεώσουμε. Αν όχι, μπορούμε να περιμένουμε. Τέλος, συμφωνώ με τα σχόλια που, έκαναν, που έκανε ο Αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου, ο κ. Μαρτίνες Μαρτίνες και συμφωνώ με τον κύριο Μαυρομάτη αν ο διαμεσολαβητή ε, σε ένα θέμα, έχει εκδώσει συστάσει, θα πρέπει πραγματικά να έχουμε πάρα πολύ ε, στεναρά επιχειρήματα για να μην δεχτούμε αυτές τις συστάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να υποστηρίξουμε το διαμεσολαβητή. Ε, βάζω εδώ απλώς ένα μικρό ερωτηματικό. Πόσο επίγον δηλαδή είναι αυτό το θέμα, αυτή η έκθεση. Ε, ε, Ευχαριστώ, κύριε θα δώσω το λόγο στον καθηγητή Διαμαντούρο για να απαντήσει σε αυτά τα ερωτήματα και συνεχεία να προσπαθήσω να συνοψίσω τη συζήτηση. Ο κύριος Διαμαντούρος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σύντομα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μαρτίνες Μαρτίνες και τον κύριο Μαυρομάτη για την υποστήριξή τους. Θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρατήρηση τώρα προς την Κομισιόν. Είναι, υπάρχει ένα θέμα ως προς την εξουσία του καθενός μας. Η Κομισιόν επέλεξε να αγνοήσει το γεγονός ότι η απόφαση του δικαστηρίου αφορά τη διαδικασία και όχι την ουσία. Μια και η ουσία ποτέ δεν εξετάστηκε και ποτέ δεν τέθηκε καν θέμα ως προς την ουσία από την Κομισιόν, Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στη δική σας θέση και στη δική μας. Το θέμα δεν είναι ότι το δικαστήριο ακύρωσε και ανέτρεψε την απόφαση του πρωτοδικίου. Το έκανε, αλλά μην ξεχνάμε ότι ποτέ δεν μπήκε στην ουσία του θέματος. Η ουσία παραμένει λοιπόν, τα επιχειρήματα παραμένουν. Αυτό που, τα ερωτήματα τώρα που έθεσε ο Σερ Ρόμπερτ. Ας απαντήσω. Μάλιστα. Φτάνει γοργά τα 65. Δεν ξέρω αν θα ήθελε να γίνει freelance διερμηνέας. Ε, ας αποφασίσει μόνος του. Καταρχάς, ε, διαδικασία έναντι ουσίας. Όπως είπα και στην Κομισιόν σε Ρόμπερτ, πιστεύω ότι αυτό που είναι ουσιώδες αυτήν την υπόθεση είναι ότι η Κομισιόν επέλεξε να επικαλεστεί την απόφαση του δικαστηρίου, του ΔΕΚ, που ακύρωνε, ανέτρεπε την απόφαση του πρωτοδικίου για διαδικαστικούς λόγους. Είπε δηλαδή ότι είναι μη παραδεκτό το αίτημα. Δεν κοίταξε ποτέ την ουσία το δικαστήριο. Επομένως η ουσία παραμένει βάσιμη. Αυτή την ουσία τη δέχτηκε το Κοινοβούλιο, η Κοινωνική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν ε, ήταν σωστό που το Κοινοβούλιο πήρε την απόφαση που πήρε, αλλά η Κομισιόν επέλεξε να μην πάρει την ίδια απόφαση. Υπάρχει και θέμα λοιπόν α, ουσίας της απόφασης του πρωτοδικίου, η οποία παραμένει. Κάτι άλλο. Γιατί μόνο οι διαρμηνείς ACI, μόνο αυτοί δεν προσλαμβάνονται. Οι βοηθητικοί υπάλληλοι είναι μια ομάδα υπαλλήλων που χρησιμοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες. Τις χρησιμοποιεί και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν μόνιμες ανάγκες και έκτακτες ανάγκες. Και το βοηθητικό προσωπικό καλύπτει τις έκτακτες ανάγκες. Η θέση μου είναι ότι το Κοινοβούλιο δέχτηκε την ιδέα ότι μπορεί κανεί να χρησιμοποιήσει αυτού του ανθρώπου ανάλογα με τι ανάγκε, ενώ η Κομισιόν λέει ότι ποτέ κανεί δεν πρέπει να του χρησιμοποιεί. Εκείνη τουλάχιστον. Τρίτον, το ερώτημα περί κακοδιαχείριση. Η κακοδιαχείριση προκύπτει από το γεγονό ότι η Κομισιόν λέει ότι για νομικού λόγου δεν μπορεί να αναλάβει δράση στο θέμα δεν δέχεται ότι μπορεί να επιλέξει να δράσει διαφορετικά. Αρνείται να δράσει διαφορετικά. Επικαλείται νομικές υποχρεώσεις και ανυπέβλητα εμπόδια. Αυτό ακριβώς συνιστά, κατά την απόψή μου, κακοδιαχείριση. Τέλος, το ερώτημά σας για το κατά πόσον είναι επίγουσα αυτή η αναφορά. Είναι δύσκολο αυτό το ερώτημα, δεν μπορώ να σας τα απαντήσω εγώ εύκολα, γιατί αυτή τη στιγμή κλείσω την έκθεσή μου εγώ, το θέμα πάει στο κυρίαρχο σώμα σας. Το σώμα σας θα αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει μια ειδική έκθεση του διαμεσολαβητή. Δεν μπορώ να σε επιβάλλω εγώ τον επίγοντα χαρακτήρα της ειδική έκθεσης. Βεβαίως, εμένα θα μου άρεσε αν τα θέματα αυτά αντιμετωπίζονται επί της αρχής και αντιμετωπίζονται με μια γρηγοράδα. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα πάρω εγώ την απόφαση, θα σα υποκαταστήσω εγώ. Εσεί θα αποφασίσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Διαμαντούρε. Ευχαριστούμε τον Ευρωπαίο Διαμασολαβητή για την απάντηση αυτών των ερωτημάτων και για την ιδιαίτερω λεπτομεριακή παρουσίαση. Ο κύριος Μαρτίνε θέλει να πάρει το λόγο ως εισηγητή Α, τρεις έλαβαν το λόγο, ο κύριος Μαρτίνεθ, ο κύριος Μαυρομάτης και ο κύριος Διαμαντούρος μέχρι στιγμής. Όλοι οι ομιλητές αναγνώρισαν ότι η παρούσα λύση από την Επιτροπή δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Και όλοι εξέφρασαν την άποψη ότι η θετική, θα πρέπει να επιζητήσουμε το ταχύτερο δυνατό μια θετική λύση. Γι' αυτό προτείνω εκ μέρους της Επιτροφής, Επιτροπής Αναφορών να επιφορτιστώ να αποστείλω, να συντάξω να αποστείλω μία επιστολή προς τον κύριο Πέτερινγκ με την παράκληση να συμφωνήσει, να εγκρίνει την προπαρασκευή αυτής της έκθεσης και να συζητηθεί η έκθεση αυτή κατά τη διάρκεια αυτής της θητείας. Δεν θα τον βάλουμε λοιπόν για την συνεδρίαση των συντονιστών νομίζω ότι θα πρέπει να πετύχουμε μια συνεννόηση μεταξύ μας ως Επιτροπή. Εάν κατάλαβα καλά τα όσα είπε ο κύριος Διαμαντούρος, ήταν ιδιαίτερος προσεκτικός και πέρασε το, ανέθεσε την ευθύνη στην Επιτροπή όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Εγώ δεν ε, έχω ξεκαθαρή άποψη όσον αφορά τον έκτακτο χαρακτήρα. Ε, δεν θέλω να αναβάλλετε μία απόφαση και έχουμε πάρει μία απόφαση στην ομάδα των συντονιστών ότι δεν θα υπάρξουν άλλες ε, εκθέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έπρεπε να προσπαθήσουμε να το κάνουμε. Και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αντιπρόεδρο, εάν θέλει αυτός να σχολιάσει για τον έκτακτο χαρακτήρα, τον επίγοντα χαρακτήρα. Εάν ε, θεωρήσει ότι είναι επίγον, εγώ θα συμφωνήσω μαζί του. Αλλά ε, μιλούμε για να το αναβάλουμε μόνο για μετά τις εκλογές, όχι για να το παραπέψουμε στις καλένδες, ε, παορίστο. Και θα εκτιμούσα πραγματικά πάρα πολύ να μας δώσει ο κύριος Μαρτίνεφ τη δική του γνώμη. Ναι, επιτρέψατε μου να σας επισημάνω ότι ο εκπρόσωπος της Επιτροπής επίσης μας ε, πρότεινε να επενεξετάσει το θέμα της Επιτροπής μελλοντικά, την άποψη της Επιτροπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ κύριε Ρόμπερτ. Εάν θέλετε να είμαι ειλικρινής, θα πρέπει να πω ότι εκτιμώ την προσέγγιση της Επιτροπής, η οποία μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει ένα πεδίο ε, συνεννόησης και νομίζω ότι θα πρέπει πραγματικά να δράξουμε αυτή την ευκαιρία, τη στιγμή ακριβώ που εκφράζεται τώρα δηλαδή. Το θέμα δεν είναι μόνο να αναβρεθεί για μετά τις εκλογές, γιατί εφόσον θα συσταθεί εκ νέου το σώμα, και εφόσον θα επανεκλεγεί ο ίδιος ο διαμεσολαβητής ή θα έχουμε ένα νέο διαμεσολαβητή. Άρα λοιπόν πάμε πολύ μακριά. Αλλά επιτρέψατε μου να είμαι ειλικρινής. Εγώ εκτιμώ πάρα πολύ τα όσα είπε η Επιτροπή, αλλά δεν θα ήμουν ειλικρινής απέναντι στην Επιτροπή ή έντιμος απέναντι στους συναδέλφους, εάν δεν έλεγα ότι υπήρξε μέχρι τώρα στεναρή μου πεποίθηση ότι η Επιτροπή θέλει να καθυστερήσει όσο μπορεί αυτό το θέμα, την επίλυση αυτού του θέματος. Ε, αυτή την εντύπωση σχημάτισε, ενδεχομένω να πατώμα, αλλά αυτή είναι η εντύπωσή μου, αυτή είναι η αίσθηση που είχα. Υπήρξε παρέμβαση, δεν ξέρω εκ μέρους ποιου, ε, προκειμένου να καθυστερηθεί το θέμα, να βρεθεί όσο γίνεται περισσότερο. Δεν ξέρω, ενδεχομένω να πατώμε και αν απατώμε ε, το θέμα είναι ξεκάθαρο. Ας ε, συνταχθεί αυτή η έκθεση ως εξαίρεση, γιατί αποτελεί μια εξαίρεση. Και ας ε, υποβάλουμε ε, σε μια δοκιμή, σε μια εξέταση την καλή θέληση, την καλή προαίρεση της Επιτροπής και θα είμαστε όλοι ευτυχείς εάν ε, η Επιτροπή φανεί συνεπής με τα όσα είπε ο εκπρόσωπός της κλείνοντας την παρέμβασή του. Πρόεδρος, Κυρίες και κύριοι, έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών. Ε, ίσως ε, αν δεν διαφωνείτε μπορώ να δώσω το λόγο στον κύριο Χάμερστάιν δεν θα ήθελα όμως να ξεκινήσει εκ νέου η συζήτηση λυπάμαι είχε κλείσει ο κατάλογος ε, των ερωτώντων όταν ε, ζήτησε το λόγο λυπάμαι δεν γίνεται να λάβει το λόγο Εσείς ήρθατε εκ των υστέρων, αφού είχα κλείσει τον κατάλογο των μιλητών. Αυτό ισχύει και για τον κύριο Χάμερσταν Μίντς. Εμείς είχαμε κλείσει νωρίτερα τον κατάλογο των ομιλητών. Άλλος παρακαλώ, ε, επιθυμεί κανείς άλλος να λάβει το λόγο, ο κύριε Ντόμπολη και ο κύριος Χάμερσταν Μίντς, μήπως και κανένα άλλος. Δεν ξέρω. Άλλος παρακαλώ, επιθυμεί κανένας άλλος το λόγο πέρα από τους ε, δύο συναδέλφους εφόσον πρόκειται για τους δύο αυτούς, εντάξει ας μιλήσω ο καθένας από 1,5 λεπτό. Αλλά λυπάμαι πάρα πολύ, ε, κατ' ουσίαν έχουμε κλείσει τη συζήτηση. Τέλος πάντων, τώρα τι γίνεται, ξαφνικά θέλουν όλοι να λάβουν το λόγο, τώρα που έκλεισε ο κατάλογος των ομιλητών. Λυπάμαι πολύ, δεν θα το καταφέρουμε από πλευρά χρόνου ας πάμε σημείο υπαριθμών 6 τη ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για την αναφορά 620 που κατέθεσε ο κύριος Στάνιεκ. Δεν ξέρω, είναι στην αίθουσα ο κύριος Στάνιεκ, είναι παρόν. Αγαπητοί κυρίε και κύριοι, διακόπτει ο πρόεδρος. Μπορείτε να μιλήσετε αν θέλετε πολωνικά να μιλήσετε στη μητρική σας γλώσσα. Έχουμε ταυτόχρονη διερμηνία. Και δεύτερον, θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Διαμαντούρου. Με συγχωρείτε, το ξέχασα αυτό προηγουμένω, κύριε Διαμαντούρε. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ευχαριστώ. E, Κύριε Στάνιεκ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητά μέλη της ε, Επιτροπής, πριν λοιπόν αποφασίσετε για το ε, κατά πόσον ε, εγκρίνεται αυτή, συμφωνείτε με αυτή την θα ήθελα να σας παρακαλέσω να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα. Γιατί μειώθηκε ο ε, πληθυσμός ε, αυτής της ε, περιοχής από 150 130.000. Το ίδιο πρόκειται η περιοχή Ζάλτσε. Το ίδιο ισχύει και για τον ε, αριθμό των παιδιών ε, στα σχολεία, από 20.000 μειώθηκε σε 2 και γιατί μιλάνε στην περιοχή αυτή τσεχικά και όχι πολωνικά. Αν τελικά το θέμα αυτό ε, παραπεμφθεί σε άλλη επιτροπή που θα κριθεί αρμόδια, θα ήθελα να κάνω το εξής ερώτημα. Η τσεχική δημοκρατία, η οποία πολλές φορές παρουσιάζεται ως τιμητής των εκθέσεων που παραπέμπονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Τι έχει να πει σχετικά με αυτά που συμβαίνουν με αυτήν την μειονότητα. Και μια άλλη ερώτηση. Ε, σύμφωνα με το άρθρο 18 της ε, Συμφωνίας Πλαίσιο για την Προστασία των ε, Μειονοτήτων, οι μειονότητες ε, έχουν δικαίωμα να απολαύουν δικαιώματα. Θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ίση προς ίσον οι κάτοικοι μιας χώρας και ε, ας μην ξεχνάμε ότι έχουμε στείλει και μία αναφορά στο Συμβούλιο της Ευρώπης όπου προτείνεται να αναστηθεί μια λύση και να εξευρεθούν και τα μέτρα ελέγχου. Και κάτι άλλο τελευταίο. Τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε ε, σχετικά με αυτήν την αναφορά. Ο ε, συνάδελφος ε, μπορεί να σας παρουσιάσει κάποια παραδείγματα για την προστασία των μειονοτήτων στην Τσεχία. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ σημαντικό και περίπλοκο ως ε, πολίτης ε, της ε, Τσεχίας αλλά με πολωνική προέλευση εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι μηχανισμοί για την αξιολόγηση και τον έλεγχο του, της εφαρμογής του χάρτη μειονοτήτων και άλλων διατάξεων της Συμφωνίας Πλαίσιο γνωρίζουμε πολύ καλά ότι όλα αυτά δεν γίνονται σεβαστά στην σύσταση 2000, του 2006 2 σε αυτή τη σύσταση ήδη έγινε η πρόταση να υπάρξουν επιτροπές μειονοτήτων έτσι ώστε οι μειονότητες να μπορούν να πτύξουν κάποιες δραστηριότητες. Και στο θέμα της ε, διγλωσίας η απόφαση για το θέμα αυτό αναβλήθηκε και ένα άλλο αδιαμφίστο γεγονός είναι το θέμα της παιδείας, της σχολικής παιδείας, όπου πράγματι υπάρχει πρόβλημα. Και κάτι άλλο, ε, το Τσεχικό Κοινοβούλιο μέχρι τώρα δεν έχει θεσπίσει καμία νομοθετική διάταξη ε, κατά της διακριτικής μεταχείρισης μειονοτήτων. Να προσθέσω ότι η Τσέχοι στην περιοχή μας δεν είναι αυτόχθονες. Προσεχώρησαν αργότερα. Ήρθαν και καταστάθηκαν στην περιοχή μας και δεν είναι ενημερωμένοι για τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ούτε καν και τα Υπουργεία της ε, Τσεχίας δεν γνωρίζουν ότι το διεθνές δίκαιο υπερισχύει του εθνικού δικαίου. Η επικύρωση του χάρτη περί γλωσσών μειονοτήτων η επικύρωση αυτή δεν έλαβε χώρα. Και επισημάνθηκε ότι πρέπει να ενισχυθεί ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης. Όμως ε, ε, τα μέσα ενημέρωση, ξέρετε, αυτά που σας παρουσιάζω εγώ τώρα, τα αποκρύπτουν. Η σύμβαση περί γλωσσών μειονοτήτων, η σύμβαση αυτή, όπως σας είπα, δεν γίνεται σεβαστή στην τσεχική δημοκρατία. Αυτά είναι ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα που ήθελα να σε αναφέρω για να τεκμηριώσω αυτά που είπε ο συνάδελφός μου. Και θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε πολύ προσεκτικά ε, όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται σε αυτή την ε, περιοχή της ε, Τσεχίας. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ότι ήρθατε εδώ και τώρα θα ήθελα να δώσω τον ε, λόγο στην Επιτροπή για να τοποθετηθεί επί του θέματος. Ο κύριος Λαδεντζάτος, ευχαριστώ. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων των ε, μειονοτήτων και ο σεβασμός της αρχής της μη διάκρισης είναι βασικές αρχές ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σεβασμός της ε, πολιτιστικής και γλωσσικής επικλημορφίας είναι ο ακρογωνιαίος λήθος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι το άρθρο 22 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, αναφέρει ότι η Ένωση σέβεται την ε, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτιστική ποικιλομορφία. Σύμφωνα με το άρθρο 51 της ίδιας της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που μιλά για το πεδίο εφαρμογής αυτών δικαιωμάτων, οι διατάξεις της χάρτας ε, ισχύουν με σεβασμό όμως της αρχής της επικουρικότητας ε, για τα κράτη-μέλη. Επομένως, αν γίνεται, γίνονται σεβαστές αυτές οι αρχές, ε, αλλά στο επίπεδο ο καθένας του τις εφαρμόζει. Σε καμία περίπτωση η χάρτα δεν τροποποιεί τις αρμοδιότητες των συνθήκων. Με βάση τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει δεσμευτική διάταξη στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτω ώστε η Κομισιόν να μπορέσει να παρέμβει στους τομείς που ανέφεραν οι αναφέροντες. Δεν μπορεί δηλαδή να κάνει τίποτα δια της δικαστικής οδού. Θα ήθελα λοιπόν να σα μιλήσω για κάποιε ουσιαστικέ πολιτικέ αρχέ που εφαρμόζει η Κομισιόν σε ό,τι αφορά την πολυγλωσία. Ε, μία αρχή που σέβεται η Κομισιόν η πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την πολυγλωσία είναι να σέβεται και τις μειωτικέ ε, γλώσσε. Το Σεπτέμβριο του 2008 στην ανακοίνωσή τη, στο κείμενο 2566 η Κομισιόν λέει ότι οι γλώσσες αυτές ε, προσθέτουν ε, μία άλλη διάσταση στην κοινή πολιτιστική μας ταυτότητα και βοηθούν στο σεβασμό των απόψεων και στην πρόθεση του διαλόγου. Όμως τα κράτη-μέλη είναι αρμόδια για την γλωσσική πολιτική ε, και για τις περιφερειακές και μειονοτικές γλώσσες. Η χάρτα για τις ε, μειωτικές γλώσσες ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης προβλέπει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο το οποίο πρέπει όλοι να σεβαστούμε. Στην ε, προηγούμενη ανακοίνωση του 2005 η Κομισιόν είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν εθνικά σχέδια με σκοπό να προωθήσουν την πολυγλωσσία, Να λάβουν υπόψη την εκπαίδευση, δηλαδή δυνατότητα εκπαίδευση των μειωτικών γλωσσών. Με βάση τα άρθρα 149, 150 και 151 της συνθήκης, τα κράτη-μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για το περιεχόμενο της ε, εκπαίδευσης και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και για την πολιτιστική και γλωσσική ε, πολυμορφία. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν ε, σκοπεύει να υποκαταστήσει τα κράτη-μέλη, αλλά να τα βοηθήσει και να τα συμπληρώσει. Τα εργαλεία που έχει η Ένωση στη διάθεσή της είναι προγράμματα χρηματοδότησης και κυρίως ε, το πρόγραμμα Lifelong Learning από το 2007 μέχρι το 2013 που δίνει ε, πολλές δυνατότητε χρηματοδότησης μέσω υποπρογραμμάτων όπως το Erasmus, ε, Leonardo da Vinci και Ludwig καθώς και διάφορες δραστηριότητε για τις γλώσσες που δίνει τη δυνατότητα επιχορήγησης σε προγράμματα και σε δίκτυα. Η Κομισιόν είναι υπέρ της εφαρμογής του διεθνούς δικαίου αλλά δεν έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί σε ένα διεθνέ δικαστήριο σε περίπτωση που δεν γίνονται σεβαστά όλα αυτά από τα κράτη-μέλη. Επομένω, αυτό το θέμα παραμένει αρμοδιότητα ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, σε νομικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο η Κομισιόν συνεχίζει τη δράση της όπως σας προανέφερα. Dziękuję bardzo. Ε, Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Στανόκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως διαβάζω σε αυτή την ε, σύσταση, που αφορά την ενημέρωση της Επιτροπής ε, ε, Πολιτικών Δικαιωμάτων και της Επιτροπής Μειονοτήτων. Θα ήθελα να πω ότι είμαι μέλος και των δύο και αντιπρόεδρος αυτού του Intergroup για τις εθνωτικές μειονότητες. Και γνωρίζουμε όλοι ότι στο πλαίσιο της ε, διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το ποσοστό των ε, παραδοσιακών ε, μειονοτήτων έχει τριπλασιαστεί. Και αυτό το θέμα είναι ιδιαίτερος ε, σημαντικό. Και ε, επίσης ε, επηρεάζει και τα παλαιά μέλη που έχουν πολλούς πρόσφυγες και έχουμε μία αναφορά σε σχέση με τα δικαιώματα ανθρώπων που έχουν εγκαταλείψει αυτά τα εδάφη εδώ και πολλούς αιώνες και έχουν και μέσω της προσέγγισης του Intergroup όσον αφορά τις εξελίξεις στην νομοθεσία όσον αφορά τη μη διάκριση έναντι των δικαιωμάτων των μειονοτήτων οι κατηγορίες αυτές θα πρέπει να διαχωριστούν και κατά την άποψή μας εθνοτικές και γλωσσικές μειονότητες, παραδοσιακές εθνοτικές και γλωσσικέ θα πρέπει να έχουν περισσότερα προνόμια, έστω και αν δεχόμαστε ότι και άλλες μειονότητες δεν θα πρέπει να εφίστανται διακρίσεις. Όσον αφορά αυτή τη σύμβαση πλαίσιο, οι χώρες έχουν κάποιες επιφυλάξεις εν σχέση με το ποιες μειονότητες αναγνωρίζουν. Η Τσεχία από όσο γνωρίζω δεν έχει τέτοιου είδους ε, επιφυλάξει όσον αφορά προσχώρηση σε αυτή τη σύμβαση. Χορηγεί λοιπόν αυτά τα δικαιώματα σε όλες τις ε, μειονότητες που ζουν στην επικράτειά της. Δε ρωτώ ε, Γιατί ε, υπάρχει αυτή η κατάσταση βεβαίω είμαστε δεθμένοι να παράσχουμε αυτές τις πληροφορίες. Είμαστε ενήμεροι ότι κατά τη διάρκεια τεσσάρων ετών των εργασιών του Intergroup και πραγματικά εξετάσαμε πάρα πολλές περιπτώσεις ιδιαίτερων ειδικών μειονοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε επίγνωση της κατάστασης και των προβλημάτων αυτών των μειονοτήτων. Γι' αυτό θεωρώ ότι οι αναφέροντες επιθυμούν μία ξεκάθαρη απάντηση εκ μέρους μας. Όχι μία απλή ενημέρωση. Μία ενημέρωση ότι αυτή η σύμβαση πλαίσιο δεν ε, ε, αποτελεί ε, κοινοτική νομοθεσία. Δεν έχει νόημα να το πούμε αυτό στους αναφέροντες. Το γνωρίζουν πολύ καλά. Το πρόβλημα είναι ε, σε ποιο βαθμό προτίθεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει ένα θετικό παράδειγμα προς όλες τις ε, χώρες μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης όσον αφορά την εφαρμογή των άρθρων αυτής της σύμβασης πλαίσιο. Και όπως είπαμε ε, δεν γίνεται κάτι τέτοιο, δεν ισχύει στην Τσεχία όπου υπάρχουν ε, κυρίως ε, πολωνικές γλωσσικές μειονότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και τη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Και νομίζω το πρώτο βήμα θα είναι να προσχωρήσει και σε αυτή τη σύμβαση πλαίσιο για τις μειονότητες η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν συνεπώς να σκεφτούμε τι είδους υποχρεώσεις θα πρέπει να αναλάβουν οι χώρες μέλη αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν γέννη εφαρμόζοντας ακριβώς αυτούς τους κανόνες του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και θα πρέπει να αναφερθώ σε αρκετά ψηφίσματα τα οποία ενεκρίθησαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου απευθύνουμε τη σύσταση προς όλες τις χώρες μέλη για παράδειγμα στρατηγικές της μη διακριτικής μεταχείρισης ένα ψήφισμα που συνέταξε η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και η Επιτροπή Απασχόλησης σε σχέση με τα δικαιώματα των μειονοτήτων και, της ακατάργησης των δια... και... και με την κατάργηση των διακρίσεων. Υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα ψηφίσματα αυτού του Κοινοβουλίου που ενεκρίθησαν από αυτό το Κοινοβούλιο και που αναφέρονται στην αναγκαιότητα που υπάρχει οι χώρες ε, μέλη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα πρέπει οι χώρες μέλη να αναστείλουν όλα τα περιοριστικά μέτρα, τους περιοριστικούς όρους που επιβάλλουν σε αυτή τη σύμβαση. Νομίζω ότι η Επιστροπή σφάλει όταν λέει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Η Δημοκρατία της Τσεχίας καθώς και η Πολωνία είναι νέα μέλη και γνωρίζουμε ότι υποχρέωση του σεβασμού των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και υποχρέωση για την κατάργηση των διακρίσεων αποτελούν τμήμα των κριτηρίων της Κοπενχάγης. Και υπό την έννοια αυτή μπορούμε να κρίνουμε τη συμπεριφορά των αρχών της Τσεχίας. η Επιτροπή ε, δέχθηκε την υποψηφιότητα της Τσεχίας. Είχε δεχτεί στο παρελθόν την υποψηφιότητα της Τσεχίας με τον όρο ότι θα πληρούνται τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Αυτό ήταν ο όρος για την προσχώρηση της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνεπώς θα πρέπει να πληρούνται αυτά τα κριτήρια. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν δύο μέτρα και σταθμά. Ευχαριστώ. Είναι παραδεκτή αυτή η αίτηση, αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ να τη συζητάμε. Οι δύο επόμενοι ομιλητές, δύο είναι, ο κύριο Τούκα Ζουόλνη και μετά η κυρία Στανισεύσκα. Ε, Πρόεδρε, Συμφωνώ με αυτά που είπαν οι εκπρόσωποι της Πολωνίας στην Επιτροπή μας. Αυτό το θέμα είναι πολύ σημαντικό. Το θέμα αυτό, αυτή τη σύμβαση πλαίσιο την έχουμε ξανασυζητήσει και είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο το οποίο έχει θεσπιστεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο και ελέγχει την εφαρμογή της ε, σύμβασης. Ε, ξέρετε ακριβώς σημαίνει η αρμόδια επιτροπή αναφέρεται στην κυβέρνηση της χώρας, η κυβέρνηση ε, και αυτή με τη σειρά της διαβάζει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή. Ε, και ακριβώς εδώ δημιουργείται το πρόβλημα, διότι οι μειονότητες δυστυχώς δεν έχουν τη δυνατότητα να παρέμβουν. Ε, παράδειγμα είναι και η Σλοβακία. Ο χάρτης περί μειονοτήτων ελέγχεται από την κυβέρνηση για το κατά πόσον ε, ισχύει και εφαρμόζεται στην πράξη, η χάρτα αυτή όχι. Όσον αφορά τη μητρική γλώσσα, η πολωνική μειονότητα στην Τσεχία, στην περίπτωση αυτή η Πολωνία θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επισημάνει τα δικαιώματα των Πολωνών στην Τσεχία. Και κατ' ουσίαν αυτό ισχύει για όλες τις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προλαλήσασα έχει δίκιο. Μετά την ένταξη αυξήθηκε κατά πολύ ο αριθμός των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε 60 εκατομμύρια 60 εκατομμύρια που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ε, μειονότητες. Στο σημείο αυτό λοιπόν θα πρέπει να επαναλάβω ότι το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει θεσπίσει πολύ σημαντικές ε, διατάξεις ε, για την χάρτα των μειονοτήτων, υπάρχει ο χάρτης ε, αυτονομίας και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα υιοθετήσουμε αυτά, έστω και με κάποιες τροποποίησεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπορεί να προσφέρει ουσιαστική προστασία των μειονοτήτων και το θέμα δεν ολοκληρώνεται με το να λέμε απλά υπάρχει η προστασία. Μα ποιο είναι το νομικό πλαίσιο στο οποίο αναφερόμεθα. Γι' αυτό λοιπόν η σύσταση την οποία έχουμε μπροστά μας ε, είναι σωστή. Βεβαίως και ευχαριστούμε που το θέμα μπήκε στην ημερήσια διάταξη και ασχολήθηκε η Επιτροπή με το θέμα αυτό. Και, και η Intergroup Παρεμπιπτόντως είμαι και εγώ μέλος της ε, Intergroup. Εδώ υπάρχει ε, κάτι το ενδιαφέρον. Το γεγονός ε, ότι η σύμβαση πλαίσιο είναι νομικό εργαλείο του Συμβουλίου της Ευρώπης που σημαίνει καταρχήν το Συμβουλίο της Ευρώπης θα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα κυρίως με, τον, με το κατά πόσον ισχύει αυτή, αυτός ο χάρτης στην πρακτική του εφαρμογή και ε, κατά πόσον ίσως ε, θα πρέπει να ρωτηθούν και οι μειονότητες αν είναι ευχαριστημένες με την εφαρμογή του χάρτη όχι. Πολύ σωστά λοιπόν οι μειονότητες αναφέρθηκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γιατί ε, όλοι οι πολίτες της ε, Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης αν κάτι ε, δεν τους αρέσει μπορούν να φερθούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το να τους στηρίξουμε και όσον αφορά την προστασία των κοινοτήτων, των μειονοτήτων με συγχωρείτε, εκεί υπάρχει κάτι στο οποίο θα μπορεί κανείς να αναφέρεται όσον αφορά την προστασία, αλλά ακόμα δυστυχώς δεν έχει εγκριθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ λίγο. Εγώ ζω 30 χιλιόμετρα από την εν λόγω περιοχή και επιβεβαιώνω αυτά που είπαν οι κύριοι που μίλησαν πριν από μένα. Έχουμε την ε, πολωνική ε, μειονότητα που ζει εδώ και αιώνες ε, στην περιοχή αυτή σε μια ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση. Και εγώ στηρίζω και αυτά που είπε και η κυρία Σδανόκα. Πράγματι πρέπει να κάνουμε τα να λάβουμε τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η Κομισιόν να προτείνει ε, συγκεκριμένες ε, νομικής φύσεως ε, λύσεις για την προστασία των μειονοτήτων, των εθνοτήτων. Σε πάρα πολλές χώρες πράγματι ισχύει αυτό η μειονότητα ε, θα το πω πολύ ήπια, δεν λαμβάνεται καν υπόψη από την πλειοψηφία. Μάλιστα, μερικές φορές υπάρχουν και κάποιες ενδείξεις διακριτικής μεταχείρισης. Μα αν δεν ασχοληθεί η πλειοψηφία για τη μειονότητα, τότε ποιος θα το κάνει. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε από την Κομισιόν να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις. Από την άλλη βέβαια, όπως σας είπα, από την άλλη βέβαια, λόγω των ε, κριτηρίων της ε, Κοπενχάγης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρέπει να υποβάλει και ένα ερώτημα προς την κυβέρνηση της Τσεχίας. Τουλάχιστον να δείξει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ανησυχεί για το πώς συμπεριφέρονται οι τσεχικές αρχές απέναντι στην πολωνική μειονότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, πράγματι θα πρέπει να αναφερθούμε στην Ευρωπαϊκή Επίτροπη με την ε, παράκληση αυτή να αναφερθεί στην ε, Τσεχία, στην κυβέρνηση της Τσεχίας, αλλά και στη μόνιμη αντιπροσωπεία της Τσεχίας και να τους ενημερώσει ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα. Κυρίες και κύριοι, νομίζω τώρα ας προχωρήσουμε πιο κάτω, ας αφήσουμε κάπως ανοιχτή αυτή την αναφορά. Ε, θα γίνει ε, μια ανακοίνωση σχετικά με το θέμα αυτό στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και θέλω να δεχθώ την πρότασή σας. Επαναλαμβάνω λοιπόν γιατί δεν άκουγε η κυρία η συνάδελφος, ε, όμως μίλησε προηγουμένως. Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Θα ε, απευθυνθούμε στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και στην Intergroup που είναι η διακομματική ομάδα εξάλλου θα έρθουμε σε επαφή και με τη μόνιμη αντιπροσωπεία της ε, Τσεχίας και θα ε, αναζητήσουμε την επαφή και με την πολωνική μόνιμη αντιπροσωπεία. Η κυρία Στανισέσκα ίσως να μην συμφωνεί απόλυτα, αλλά εγώ νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να δραστηριοποιηθεί κυρίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα, ε, όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να επεξεργαστεί ένα φάκελο όσον αφορά το θέμα αυτό. Πρόεδρε, θα ήθελα να αλλάξουμε λιγάκι τη διατύπωση. Γιατί ε, να αναφέρεται ότι θα αναζητήσουμε περισσότερο ε, την έρευνα του θέματος από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και όχι απλά την ενημέρωση. Εντάξει, σύμφωνα. Ω εκ τούτου κλείνουμε αυτό το σημείο της σημερινής διάταξης. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Στάνιεκ και τον ε, σύνοδό του. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και θα σας ε, συνεχίσουμε να σε ενημερώνουμε για τη συνέχεια της υπόθεσης. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας ανακοινώσω ότι ο κύριος Κάστλερ είναι το νέο μέλος της Επιτροπής μας που προέρχεται από το ΕΛΚ. Σας καλωσορίζω θερμά. Προχωράμε. Πάμε στο σημείο υπαριθμών 7 τη ημερήσιας διάταξης. Η αναφέρουσα είναι παρούσα. Ε, πρόκειται ε, για μια διπλή αναφορά την 188 και την 1198. Πρόκειται για το ίδιο θέμα. Στην δεύτερη περίπτωση ε, ο αναφέρον είναι ο κύριος Μαγιόρ. Είστε παρόν? Είστε εδώ? Παρόν ο κύριος Μαγιόρ? Κύριος Μαγιόρ, είναι παρόν. Σπατρujemy το, το poproszę o zabranie głosu Εφόσον ο κύριος Μαγιόρ ή κάποιος εκπρόσωπός του δεν είναι εδώ, πρέπει να προχωρήσουμε, αλλά μας είχαν πει ότι θα ερχόταν. Να δώσω το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Κέστερ, Ράντι Κέστερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας παραπέμψω στην ανακοίνωση της Κομισιόν της 25ης Ιανουαρίου του 2007, γιατί η νέα αναφορά ουσιαστικά επαναλαμβάνει τα επιχειρήματα ε, μιας αναφοράς που είχε υποβληθεί το 2006. Τότε η Κομισιόν είχε έρθει σε επαφή με τις πολωνικές αρχές, ε, έλεγξε το θέμα και είχε ενημερώσει εκτεταμένα την Επιτροπή Αναφορών δεν θεωρούμε ότι υπάρχουν περιοριστικές πολιτικές ή κάποια παραβίαση του κοινοτικού δικαίου σε ό,τι αφορά την απόσπαση εργαζομένων μεταξύ Πολωνών και Γερμανών ή οποιονδήποτε άλλων ε, κρατών μελών. Έχουμε το γενικό κανόνα που αφορά τους ε, εργαζομένους και τον τόπο λειτουργία τους. Υπάρχουν εξαιρέσεις όμως για την απόσπασή τους. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συντρέχουν ορισμένες, ε, να γίνονται σεβαστές ορισμένες προϋποθέσεις για να δεχτούμε ότι πρόκειται για εξαίρεση από το γενικό κανόνα. Αυτή η προϋπόθεση, ε, οι προϋποθέσεις μάλλον, αναφέρονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και από τις αποφάσεις του 10. Ε, Επίσης, η διαδικασία έχει συγκεκριμενοποιηθεί περαιτέρω μέσω της απόφασης της Επιτροπής ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα δικαιώματα των ε, μετακινούμενων εργαζομένων. Με βάση τα στατιστικά μας δεδομένα το 2005 υπήρχαν 82.000 έντυπα ε101. Το 2006 163.000 και 120.000 από την Πολωνία στη Γερμανία. Το προηγούμενο ήταν από τη Γερμανία στην Πολωνία. Έχουμε δηλαδή μια στατιστική αύξηση αυτών των εντύπων. Η Κομισιόν δεν έχει ενημέρωση ότι υπάρχει κάποια ε, περιοριστική πολιτική, κάποια περιοριστική συμφωνία μεταξύ Γερμανίας και Πολωνίας για να παραβιάσουν τους κανόνες που ισχύουν σε αυτό το τομέα από το κοινοτικό δίκαιο και από τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Θα πρέπει να προσθέσουμε ότι αυτοί οι κανόνες για την έκδοση των εντύπων αφορούν την παραμονή σε ένα νέο ε, κράτος μέλος ε, για 12 μήνες το πολύ του εργαζόμενου. Και σκοπό έχουμε να υπάρχει, να εξασφαλίσουμε ισορροπία μεταξύ κομικής ελευθερίας και της προστασίας α, των εργαζομένων. Θέλουμε να αποφύγουμε το κοινωνικό dumping. Θα πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθε, προϋποθέσεις για την απόσπαση εργαζομένων σε ένα άλλο κράτος μέλος ούτω ώστε να μην διαταράσουμε την τοπική αγορά εργασία, δηλαδή την αγορά εργασία ενό άλλου κρατού μέλου. Σας παραπέμπω ακριβώ γι' αυτό στην ανακοίνωση της 25ης Ιανουαρίου του 2007. Ε, εκεί καταλήγουμε ότι δεν έχουμε πληροφορίες ότι οι πολωνικές αρχές ε, προβαίνουν σε κακοδιαχείριση. Ε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε για την έκδοση του πιστοποιητικού ε101. Η τάση είναι αυξητική και γίνεται ε, πληρη σεβασμός των κανόνων και των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Έχουμε ένα εκπρόσωπο της πολωνικής ε, μόνιμης ε, αντιπροσωπείας. Θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι. Εκ μέρους της πολωνικής ε, μόνιμης αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήθελα να πω δύο λόγια για τις δύο αυτές αναφορές της κυρίας Κραζούτσκα και του κύριου Μαγιόρ. Συμφωνούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το θέμα αυτό. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων έχει κάνει μια δήλωση στην Πολωνία για αυτό το θέμα, λέγοντας ότι οι πολωνικές αρχές εξέτασαν τις ε, κατηγορίες της ε, Ένωσης ε, Πολωνών Εργοδοτών και βρήκαν ότι οι πληροφορίες μεν είναι σωστές, αλλά ότι η έρευνα δεν επιβεβαίωσε σε καμία περίπτωση πρακτικές περί δωδεκάμινης διακοπής ανάμεσα σε δύο διαδοχικές αποσπάσεις μέσα σε μία πενταετή περίοδο όπως αναφέρει το άρθρο 14 του 1408 για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Θα ήθελα να σας τονίσω ότι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην Πολωνία μπορεί να επανεξετάσει χωρίς κανένα πρόβλημα την ουσία της αναφοράς εάν η Ένωση Πολωνών Εργοδοτών μπορεί να μας δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα πρακτικών που δεν ευθυγραμμίζονται με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Δεν νομίζω ότι έχω να πω τίποτα άλλο για αυτό το θέμα προς το παρόν. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Άλλος κανείς θέλει να πάρει το λόγο. Εδώ έχουμε ένα διαφορετικό πρόβλημα. Έχουμε την Ένωση Πολωνών Εργοδοτών. Και, ε, ο κύριος Μαγιόρ μας είχε πει ότι θα ερχόταν. Είμαι λίγο πρόθυμος να κλείσω αυτή την αναφορά, γιατί πραγματικά μέχρι την τελευταία στιγμή με διαβεβαίωσαν ότι θα ερχόταν στη συνεδρίαση. Και η Επιτροπή και η πολωνική κυβέρνηση έχουν τις ίδιες απόψεις για αυτό το θέμα, αλλά όμως η αναφορά από την Ένωση Πολωνών Εργοδοτών μιλάει και για το πολωνικό και για το γερμανικό σύστημα κοινωνικών ασφαλίσεων. και μιλάει για ζημία προς τους Πολωνούς εργαζομένους. Θα ήθελα να ακούσω πραγματικά τη γνώμη του κ. Μαγιόρ, γιατί άπαξ και κλείσει κανείς μία αναφορά, είναι δύσκολο να την ξανανοίξει. Γι' αυτό θα έλεγα να βάλουμε αυτή την αναφορά στον κατάλογο των αναφορών Β και αν προκύψουν νέα επιχειρήματα από τον κύριο Μαγιόρ, μπορούμε να επανεξετάσουμε αυτή την αναφορά να το κάνω αυτό επειδή λείπει σήμερα ο κύριο Μαγιόρ. Ε, δεν ξέρω αν η γραμματεία έχει να πει κάτι διαφορετικό. Όχι. Πολύ ωραία. Άρα μπορούμε να κάνουμε αυτό που σας είπα. Σας ευχαριστώ όλους. Προχωράμε τώρα στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης, αναφορά 1007 του 2006 για το Γερμανικό Στοξιδοτικό Ταμείο DRB. Ο κύριος ε, Κάστα Ρόντι Κάστρα από την Κομισιόν ξανά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα πω πολύ περισσότερα πράγματα από αυτά που έγραψα ήδη. Δύο φορές ήρθαμε σε επαφή με τον αναφέροντα. Δυστυχώς δεν ήρθε σε επαφή μαζί μας και του στείλαμε μία, ένα αντίγραφο της απόφασης του δικαστηρίου στο Ανόβερο γιατί βάσει των πληροφοριών που έχουμε λάβει από τα γερμανικά όργανα ε, μια, υπήρξε μάλλον μία δικαστική διαδικασία και ο αναφέρον δεν ήρθε σε επαφή μαζί μας, δεν μας διαβίβασε καμία σχετική πληροφορία Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ε, παραπέμψω στην ανακοίνωσή μας και θα ήθελα να σας τονίσω ότι εδώ ότι πρόκειται για μία διένεξη που αφορά ε, διακρατικές συμφωνίες και όπως φαίνεται η, ίδια, η Επιτροπή δεν είναι δυνατόν να παρέμβει στις αποφάσεις των αρμόδιων γερμανικών δικαστηρίων και σε περίπτωση που ο ετών θεωρεί ότι τα δικαιώματά του δεν έχουν ε, ληφθεί επαρκώς υπόψη ή δεν έχει υπολογιστεί σωστά η σύνταξή του στη Γερμανία υπάρχει, η μοναδική δυνατότητα είναι να προσφύγει στα αρμόδια εθνικά δικαστήρια. Δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα. Συνεπώς δεν έχω να σας δώσω άλλες ε, πληροφορίες. Ε, μπορώ μόνο να επαναλάβω ότι του γράψαμε ε, δύο φορές και δεν μας έστειλε απολύτως καμία απάντηση. Ο κύριος Μαυρομάτης έχει το λόγο. Είναι σαφής, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο καταλήγει στην ανακοίνωσή της σήμερα, στα όσα μας είπε ο εκπρόσωπό της, ότι από τη στιγμή κατά την οποία ζητήθηκε από την Κομισιόν να δει κατά πόσον στα δικαστήρια εκρεμεί, στα εθνικά δικαστήρια εκρεμεί αυτό το θέμα και απάντηση δεν υπάρχει, δύο λύσεις υπάρχουν. Πρώτον, είτε ότι υπάρχει κάποια απόφαση και την αγνοεί ο αναφέρον, είτε δεν έχει φτάσει ακόμα και επομένως κλείνει ή αφήνουμε ανοιχτή αυτή την υπόθεση. Στην περίπτωση κατά την οποία ο αναφέρον δεν ανταποκρίθηκε σε αυτό που ζήτησε η Κομισιόν σημαίνει ότι έχει τελεσιδικήσει. Άρα δεν υπάρχει λόγος να κρατούμε ανοιχτή αυτή την ε, αναφορά. Ευχαριστώ. Tak jest, ja się zgadzam z tym, także myślę, że w świetle odpowiedzi Komisji Europejskiej tych ναι, με την άποψή σας. Υπό το πρίσμα της απάντησης που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον όσον είπε ο κ. Μαυρομάτης μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό και να περάσουμε στα επόμενα σημεία της ημερής διάταξης 9, 10 και 11. Πρόκειται για παρόμοιες περιπτώσεις, πρόκειται για περιπτώσεις ασθενών που υποφέρουν από σκλήρινση κατά πλάκας. Θα ήθελα να χαιρετήσω τους αναφέροντες και να τους πω πόσο εκτιμούμε την προσωπική τους παρουσία εδώ. Η κυρία Ντρομπίνσκα παρίσταται εδώ, εάν δεν απατώμε, μάλιστα. Ε, εκπροσωπώ τον ε, Πολωνικό Σύνδεσμο των ασθενών που πάσχουν από σκλήρινση κατά πλάκας. Έχει γίνει μια σχετική συζήτηση για αυτή την ασθένεια και θα ήθελα να παρακαλέσω την εκπρόσωπο του, της Πολωνικής ε, Ένωσης ατόμων που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας να πάρει το λόγο. Η, Πολωνική, Ένωση των ασθενών αυτών υπέβαλε αυτή την αναφορά σε σχέση με την δυσμενή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι ασθενείς και τις πραγματικά ε, ελλειπείς αντιδράσεις της ε, πολωνικής ε, κυβέρνησης σε σχέση με τα εθνικά προγράμματα καταπολέμησης αυτής της νόσου. Ένα μισή χρόνος έχει περάσει από την υποβολή της ε, αναφοράς και λόγω της δημιουργικής κατάστασης των ασθενών και λόγω πολλών μέτρων που είχαν εξαγγελθεί θα μπορούσε κανείς να πιστεύει ότι το κείμενο αυτό πλέον έχει χάσει την αξία του, είναι εντελώς παροχημένο. Αλλά δεν ευσταθεί αυτό γιατί η πολωνική κυβέρνηση δεν έλαβε απολύτως κανένα μέτρο για τη βελτίωση της κατάστασης των ασθενών και συνεπώς ε, μοιάζει απολύτως δικαιολογημένος ο ισχυρισμός ότι πρόκειται εδώ για μια διάκριση εις βάρος των ασθενών αυτών όσον αφορά την ε, δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπεία και οι ε, ασθενείς αυτοί, συγγνώμη, αποκλείονται από το κοινωνικό βίο. Οι αλλαγέ στην ε, Πολωνία από την εποχή της υποβολής της αναφοράς ε, είναι ανεπαρκής. Δεν μπορεί κανείς να πει δηλαδή ότι η κατάσταση ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και σε αυτό συνηγορούν τα εξή επιχειρήματα η δυνατότητα πρόσβασης σε θεραπείες, θεραπείες που είναι ρουτίνα στην Ευρώπη ε, εξασφαλίζονται μόνο για το 3% των ασθενών. Σύμφωνα με το βαρόμετρο μιας ε, ευρωπαϊκής ε, πλατφόρμας που διενήργησε την ελόγω έρευνα καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κατάσταση αυτή στην Πολωνία είναι η χειρότερη. Η Πολωνία είναι μία από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη όπου όσον αφορά τη διάρκεια της θεραπείας και την αγωγή ε, τελικά κρίνουν ε, παράμετροι μη ιατρικοί. Ε, η αγωγή διαρκεί συνήθως τρία χρόνια, ενώ οι ειδικοί λένε ότι η αγωγή θα πρέπει να συνεχίζει όταν έχουμε το ευκταίο θεραπευτικό αποτελέσμα. Ε, τώρα, όσον αφορά τα κέντρα θεραπείας και αποκατάστασης των ασθενών, θα πρέπει να πούμε ότι είναι απολύτως ανεπαρκή. Και πέρα από αυτό υπάρχουν πολλές διαφορές όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβαση σε διάφορες θεραπευτικές μεθόδους. Στην Πολωνία η θεραπεία της νόσου αυτής και, τα, και οι απαιτήσει προς τα, προς τα κέντρα αυτά ή μάλλον το επίπεδο ε, υπηρεσιών σε αυτά τα κέντρα ποικίλουν σημαντικά και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι ασθενείς να πρέπει να αλλάζουν συχνά το από διαμονής για να μπορούν να έχουν μια πιο ποιοτική αγωγή, θεραπεία. Και εκτός τούτου δεν υπάρχει κανένα σύστημα όσον αφορά τη συμπερίληψη και μια ψυχολογικής διάσταση στη θεραπεία. ο πολωνικός εργανισμός εκπώνησε ένα εθνικό πρόγραμμα θεραπείας που προσεγγίζει την νόσο σαν μια πολύπλοκη οντότητα. Αυτό το πρόγραμμα υποβλήθηκε, το σχέδιο προγράμματος μάλλον υποβλήθηκε στην κυβέρνηση αλλά μέχρι στιγμής δεν είχαμε απολύτως καμία απάντηση τα πρόσωπα τα οποία είναι αρμόδια για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα μας αγνόησαν απολύτως τα αιτήματά μας. Ο κύριος Μάλεκ Φεντόσκι, ο υφυπουργό Υγείας, δήλωσε δημόσια ότι τα προβλήματα αυτά θα πρέπει να επιληθούν μέχρι τα τέλη του 2008, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να τηρήσει τις υποσχέσεις του λόγω ακριβώς του γεγονότος ότι τα βήματα τα οποία εξήγηλε η κυβέρνηση τελικά δεν υλοποιήθησαν στο ε, περιβάλλον των ασθενών της νόσου αυτής δεν υπάρχει απολύτως καμία ελπίδα για τυχόν βελτίωση της κατάστασης. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω το εξή. Έχετε αυτά τα στατιστικά στοιχεία στη διάθεσή σας από τα οποία μπορούμε να δούμε ποια είναι η θέση της ε, Πολωνίας. Παρακαλώ να διαβάσετε τα στοιχεία αυτά στη γραμματεία μας. Και τώρα θα ήθελα να σας προτείνω ο συντάκτης της αναφοράς να πάρει το λόγο που προβλέπεται κάτω από ένα άλλο σημείο της ημερήσιας διάταξης, το 10. Πρόκειται για τον Κάλλος Ρικέλ με θέλει. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Είναι Ισπα... Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λέγομαι Κάλλος Ρικέλ με Φελίπ. Είμαι από τη Βαρκελόνη και έχω σκλήνηση κατά πλάκας. Όταν έκανα την ε, αναφορά ήταν το 2006 και η νόσος ε, βρισκόταν υπό εξέλιξη. Και γι' αυτό λοιπόν υπέβαλα την αναφορά αυτή, αλλά δεν είμαι σε να τη διατυπώσω με την απαιτούμενη σαφήνεια. μια μεγάλη υπάρχει μια μεγάλη διαφορά μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών περιοχών όσον αφορά την προσοχή που δίνεται στους ασθενείς πάσχων από σκλήνηση κατά πλάκας. Ε, και υπάρχει μια διάκριση κατά των ασθενών βάσει ακριβώς του τόπου καταγωγής τους ή του τόπου διαμονής τους. Και πιστεύω ότι η διάκριση αυτή συνεχίζει να υπάρχει ε, και θα πρέπει να καταργηθεί. Πιστεύω επίσης ότι υπάρχει ένας ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκός κώδικας σωστής ε, συμπεριφοράς που πραγματικά θα μπορούσε να βελτιώσει την κατάσταση και να συμβάλλει στο να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπρος. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή αυτή να ασκήσει πίεση στην Ισπανική κυβέρνηση, ούτως ώστε όλες οι περιοχές της Ισπανίας, όλες οι αυτόνομες κοινότητες ε, να παρέχουν ισότιμες, ε, ισότιμες συγγνώμη, θεραπείες ούτω ώστε οι ασθενείς ολόκληρη την επικράτεια της Ισπανίας να έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν τα ίδια φάρμακα και να έχουν μια ίση πρόσβαση στις θεραπείες. Θα ήθελα να δώσουμε, να τώρα να δώσετε το λόγο στον πρόεδρο του Ισπανικού Οργανισμού για την καταπολέμηση της κλήρυνσης κατά πλάκας που είναι σε θέση να εκφράσει καλύτερα από μένα Αυτό που θέλω να πω γιατί πραγματικά δεν μπορώ, δεν είμαι σε θέση πλέον να συνεχίσω την παρέμβασή μου. Ε, ευχαριστώ πολύ Κάλλος. Εσύ στη ιδέα που εκφράστηκε εδώ πράγματι στην Ισπανία υπάρχει ένα αποκεντρωμένο σύστημα μέσω των αυτόνομων επαρχιών και ο κύριος Ρικέλμε είπε ότι δεν υπάρχει μια... σε ορισμένες περιοχές δεν υπάρχει δυνατότητα ε, πρόσβασης θεραπείες σε ορισμένες περιοχές. Ε, και αυτό όμως που συμβαίνει στην Ισπανία συμβαίνει και σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Ε, υπάρχει ευρωπαϊκός κώδικας για, την, για τις σωστές πρακτικές, αλλά νομίζω ότι δεν λαμβάνεται υπόψη ή συγκεκριμένα στην Ισπανία δεν ε, λήφθη υπόψη την εποχή εκείνη. Στην Ισπανία κάνουμε πολλές προσπάθειες ούτως ώστε να ισχύει ο κώδικας αυτός και θεωρούμε ότι θα πρέπει να γίνει σύσταση εκ μέρου τη Επιτροπή σα ή εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτω ώστε πραγματικά να εφαρμοστεί ο κώδικα αυτό. Αναφίβολα πρόκειται για ένα ζήτημα πολιτική ε, βούληση, να πετύχουν χρήματα ε, για την ασθένεια αυτή. Στη Βαρκελόνη υπάρχει πλήρη έλλειψη στατιστικών στοιχείων η κατάσταση γενικά στην Ισπανία ίσως δεν είναι τόσο κοκκή αλλά δεν έχουμε καθόλου στοιχεία και δείκτες για να γίνει μια σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει αυτός ο κώδικας σωστής συμπεριφοράς, ευρωπαϊκός κώδικας, για να μπορούν να γίνονται και αυτές οι συγκρίσεις. Ε, επαναλαμβάνω ότι υπάρχει, υπάρχουν σημαντικές ε, διαφορές μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών ε, περιοχών και θα πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο Ευρωπαϊκός Κώδικας σε σχέση με τις ε, υπάρχουσες θεραπευτικές αγωγές και τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, τα οποία είναι καλά και τα οποία θα συνεχίζουμε να χρησιμοποιούμε ώστε να καταπολεμήσουμε την επίπτωση αυτής της νόσου. Ευχαριστούμε πολύ. Εξ ονόματος της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, θα τοποθετηθεί για αυτά τα δύο θέματα ο κύριος Λουκ Φάι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ε, να παρουσιαστώ η Μονίκ Φάι από την Διεύθυνση Γενική Διεύθυνση για την Προστασία του Καταναλωτή και για θέματα υγείας που για εσωτερικούς δικούς μας διοικητικούς λόγους είναι αρμόδια και για θέματα τα οποία έχουν σχέση με όλες τις μεταδοτικές ασθένειες. Πριν λοιπόν σας παρουσιάσω την θέση της Κομισιόν, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω τις ευχές μου και την κατανόηση που έχω στους αναφέροντες. Νομίζω ότι αυτό ισχύει για όλους όσοι βρίσκονται στην αίθουσα. Και αυτό ισχύει Κυρίως για το ότι δεν είναι μόνοι τους, ε, οι πληροφορίες που έχουμε στον αφορά τη σκλήνηση κατά πλάκας ιδιαίτερα, αλλά και γενικότερα και άλλες ε, ασθένειες, είναι ότι πράγματι υπάρχει ανισότητα στη θεραπεία, ακόμα και εάν σε ολόκληρη την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν ευέλτιστες πρακτικές ή προσπάθεια προς την εφαρμογή αυτών. Είναι δύσκολο βέβαια ε, για μένα να πω οτιδήποτε άλλο ή να το εκφράσω αλλιώς το θέμα, γιατί ακόμα και το να συλλέξει κανείς στοιχεία για αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα θέματα που συγκεντρώνουμε δίνουν μια πολύ σαφή εικόνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά το θέμα και μάλιστα έχουμε στηρίξει προγράμματα κυρίως στον τομέα αυτό για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στοιχεία και πληροφορίες έτσι ώστε να κάνουμε τη σύγκριση ανάμεσα στα κράτη-μέλη και μέσα στα ίδια τα κράτη-μέλη. Και βοηθάμε στη χρηματοδότηση των προγραμμάτων που έχουν οδηγήσει στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Συμπεριφοράς όσον αφορά τη σκλήρινση κατά πλάκας, κάτι στο οποίο αναφέρθηκε ο δεύτερος κύριος που έλαβε το λόγο. Παρ' όλα αυτά, ε, νομίζω κύριε Πρόεδρε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουμε πληροφορίες που κατατείνουν στο ότι υπάρχουν ανισότητες. Υπάρχουν ξεκάθαρα σημεία αναφοράς όσον αφορά τις ε, βέλτιστες ε, πρακτικές. Αυτό δεν το λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά το συμπεραίνουμε από άτομα τα οποία εμπλέκονται με όλη αυτή την υπόθεση μέσα από επαγγελματίες, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τον τομέα. Και έχουμε λοιπόν αυτά τα σημεία αναφορά σχετικά με τις ευέλτιστες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στη τελική ανάλυση όμως κύριε Πρόεδρε, η, ε, σύμφωνα με τις συνθήκες η κατανομή των ορμοδιοτήτων και οι ευθύνες ε, καθορίζονται σε όλους τους τομείς υγείας ε, και νομίζω ότι ε, μπορώ να προσπαθήσω να εξηγήσω και αυτά που μας λέει ο αναφέρον. Η ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την υγεία ορίζεται στο άρθρο 152 της συνθήκης, της ιδρυτικής συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δικός μας λοιπόν ο ρόλος είναι να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη, πράγμα που πράττουμε, προσφέρουμε πληροφορίες, βέλτιστες πρακτικές, διευκολύνουμε τη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη, όπως επίσης και τη σύγκριση ε, με βάση κάποια συγκεκριμένα κριτήρια. Και ε, αυτό το πράττουμε βεβαίως και στον τομέα και της σκλήρινσης ε, κατά πλάκας. Το άρθρο αυτό της συνθήκης αναφέρει με απόλυτη σαφήνεια ότι πρέπει να σεβόμεθα τις αρμοδιότητες των κρατών μελών για την παραθέτω οργάνωση και παροχή ιατρικών υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Τέλος της παράθεσης. Που σημαίνει ε, χρησιμοποιώντας, ε, αν δούμε λιγάκι τι σημαίνει αυτή η γλώσσα που χρησιμοποιείται, καταλήγουμε στο ότι ε, η παροχή πληροφοριών είναι θέμα των κρατών μελών και των εθνικών και περιφερειακών αρχών για να καταλήγουν εκείνες στο τι χρηματοδοτούν, σε τι υπηρεσίες παρέχουν και ποιες όχι. καταλαβαίνουμε πολύ καλά την απογοήτευση που υπάρχει από πλευράς αναφερόντων και προσπαθήσαμε, νομίζω Πρόεδρε, στην απάντησή μας να περιγράψουμε τις διάφορες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Λυπάμαι όμως, αλλά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο πιο συγκεκριμένο σε σχέση με την υπόθεση την οποία παρουσίασαν. Πρόεδρος, ε, ευχαριστούμε πολύ. Ε, ο κύριος ε, Μαυρομάτης, ο κύριος ε, Κάσμαν, Στανισεύσκα και ακόμα ένας επιθυμεί, κάποιος άλλος το λόγο. Αν όχι, θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Τέσσερις έχουν ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να σας ε, παρακαλέσω να είσαστε σύντομοι στις ε, παρεμβάσεις σας, να μην ξεπεράσετε τον χρόνο των δύο λεπτών, γιατί ε, έχουμε και κάποια άλλα σημεία της μεσηδιάδεξης που πρέπει να εξετάσουμε παρουσία των αναφερόντων. Ο κ. Μαυρομάτης παρακαλώ. Η ηθική μας στήριξη στους πάσχοντες και όσους ακόμα βρίσκονται εδώ σήμερα, πάσχοντες από την σοβαρή αυτή ασθένεια, καθώς και τους αναφέροντες βεβαίως, στους οποίους θα πρέπει και να συμπαρασταθούμε, αλλά και να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή. Από τη δική μου πλευρά θα ήθελα να πω ότι ήδη από το 2005 αντιμετώπισα για την χώρα μου την Ελλάδα μια ανάλογη περίπτωση όπου οι πάσχοντες ήρθαν, με είδαν και είπαν για τις ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτόν τον τρόπο της θεραπείας, της αγωγής και γενικότερα για τους ανθρώπους στην ε, σκλήρηση κατά και τους ασθενείς στην Ελλάδα μέσω της Επιτροπής στην οποία μετήχα, την Επιτροπή Ανάπτυξης και τον ε, προϋπολογισμό, τότε εγκρίθηκαν με τροπολογία μου 10 εκατομμύρια ευρώ συγκεκριμένα για τους σκοπούς τους οποίους ζήτησαν οι πάσχοντες στην Ελλάδα και ο σύνδεσμος τουλάχιστον των ανθρώπων αυτών που χρειαζόντουσαν και τα χρήματα για, την περαιτέρω θεραπεία ή τις θεραπείες που είναι ήδη αναγνωρισμένες. Με πρόσφατη ερώτησή μου για το ίδιο θέμα στην Κομισιόν και χαίρομαι που εδώ αναφέρθηκαν περί προγραμμάτων η Κομισιόν υπάρχει στον προϋπολογισμό του 2007-2013 ποσό 16 δισεκατομμυρίων ευρώ για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα, την θεραπεία, την αγωγή σε όλες τις χώρες. Αυτό τι σημαίνει κύριε Πρόεδρε, ότι πρέπει να κινηθούμε όλοι και τα κράτη-μέλη και εμείς που εκπροσωπούμε τους πολίτες των 27 κρατών μελών ώστε τα χρήματα αυτά και έγκαιρα να βρίσκονται στην διάθεση των πασχόντων ή των κρατών μελών για όποιους σκοπούς χρειαστεί από εδώ και στο εξής. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι θέμα και των κυβερνήσεων να λάβουν υπόψη αυτά τα μέτρα και να μην καταγγέλουμε και κατηγορούμε πάντα την Κομισιόν ότι δεν κάνει την, ε, τη δουλειά της. Χρειαζόμαστε κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι και εμείς να συντονιστούμε και να προτρέψουμε τους κυβερνώντες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Dziękuję bardzo. Pan Kaszman, dwie minuty.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 and the best treatment that is available. Να υποβαθμίζουμε, πρέπει να αναβαθμίζουμε τη θεραπεία και γι' αυτό λοιπόν χαιρετίζω το γεγονός ότι η Κομισιόν ε, προσπαθεί να παρουσιάσει σωστές κατευθυντήριες γραμμές ε, για την ποιότητα της ε, ζωής και για την θεραπεία που προσφέρεται. Σημείωσα ότι προβλέπεται ένα συνέδριο για το 2009 το 2010 και θα ήθελα να πω στην Κομισιόν καλύτερα το συνέδριο αυτό να γίνει το 2009 και όχι το 2010 γιατί πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα το θέμα. Ε, για να ανακεφαλαιώσω λοιπόν, ε, ε, χρειαζόμαστε ελάχιστες προδιαγραφές, πρέπει να προσφέρουμε τις βέλτιστες δυνατές υπηρεσίες και το ανώτατο επίπεδο ζωής. Χρειαζόμαστε την καλή πρακτική και βεβαίως το θέμα της αρμοδιότητας των κρατών μελών, όμως είναι αρμοδιότητα των πολιτικών να υπενθυμίζουν στα κράτη-μέλη τις ευθύνες τους και να τους επισημαίνουν που ακριβώς αποτυγχάνουν. Είναι καθήκον μας αυτό και είμαι σίγουρος ότι οι αναφέροντες ε, δεν θα ε, φοβηθούν να επισημαίνουν συνέχεια αυτές τις ευθύνες. Συγγνώμη κύριε Μαυρομάτη, είχα ξεχάσει να ανοίξω το μικρόφωνο. Χίλια συγγνώμη. Πρόεδρος, ε, Μάλλον, ε, θα ήθελα να υποστηρίξω απόλυτα αυτά που είπε ο κύριος ε, Κάσμαν. Αν ε, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της την κινητικότητα και την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών, τότε αναγκαστικά αυτό οδηγεί στο ότι οι ε, συνθήκες πλαίσιο για την αντιμετώπιση ασθενειών θα πρέπει να είναι παρεμφερή στα κράτη-μέλη. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει και για τις σπουδέ. Να μπορεί κανείς να ξεκινάει σπουδέ σε ένα α κράτος μέλος, να συνεχίσει ένα β και να ολοκληρώνει σε ένα τρίτο κράτος μέλος. Βεβαίως και η παιδεία είναι αρμοδιότητα των κρατών μελών, όμως γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ξεκίνησε η, ε, συνθήκη, η εφαρμογή της συνθήκης της Μπολόνια έτσι ώστε να υπάρξει μια ομοιομορφία όσον αφορά τις ε, εκπαιδευτικές ε, συνθήκες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο ε, χρειαζόμαστε τον τομέα της υγείας και την πολιτική υγείας. Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει σαφής κοινοτική πολιτική και αυτό το επισήμανε και ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, δηλαδή δεν έχουμε μόνο το δικαίωμα αλλά και την υποχρέωση να κάνουμε σωστή ενημέρωση τότε ε, θα είχαμε και ε, τακτές ε, εκθέσεις για το πώς ακριβώς αντιμετωπίζονται οι ασθενείς στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα μπορούσαμε να έχουμε την ανάλυση δεξιοτήτων αυτό τώρα αναφέρουμε περισσότερο στο θέμα της παιδείας, τη μελέτη πίζα, της πίζα, πώς ακριβώς μπορεί κανείς να εντοπίσει τις δεξιότητες των ε, μαθητών γιατί αυτό ε, θα ήταν ένα πολύ καλό εργαλείο των ενδιαφερομένων απέναντι στο κράτος τους. Γιατί σε καθένα κράτος ε, δεν αρέσει να είναι ουραγός σε έναν κατάλογο. Ως εκ τούτου είμαι σίγουρη ότι τα κράτη-μέλη θα κατέβαλαν προσπάθεια για να ανέβουν σε ένα ενδεχόμενο κατάλογο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας ε, ιδιαίτερα αποτελεσματικός ε, μηχανισμός. Ο κύριος ε, Σάντερτς για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ επίσης θα ήθελα να εκφράσω τη δική μου αλληλεγγύη προς τους ετούντες που σήμερα μας συνοδεύουν καθώς και προς όλους τους ασθενείς που υποφέρουν από σκλήρυνση κατά πλάκας. Θεωρώ ότι, στην Ευρωπαϊκή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά να δράσει στο επίπεδο αυτό. Κυρίως όσον αφορά ε, δεδομένα αυτής της ασθένειας. Θα ήθελα να σας πω ότι ε, ένα θέμα είναι η ανισότητα και ένα άλλο ζήτημα είναι η αποκέντρωση. Θα πρέπει να μεριμνήσουμε ούτε ώστε όλοι οι πολίτες να έχουν ε, ίσων προδιαγραφών αγωγές, θεραπείες. Ο κύριος ε, Καρλ Ρικέλμε προέρχεται από την Καταλωνία και ήθελα να του πω ότι υπάρχει μια θετική βούληση τα τελευταία χρόνια όσον αφορά το πρόγραμμα υγείας και υπάρχει μια αύξηση, ένας τριπλασιασμό των πόρων για την οικία τα τελευταία τρία χρόνια, από το 2005 στο 2008 και ε, ε, ελπίζουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανταποκριθεί ε, θετικά σε αυτές τις εξελίξεις. Τώρα... Πρόεδρος, τώρα λοιπόν θα ακούσουμε την τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη σκλήνηση κατά πλάκας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να αδράξω την ευκαιρία για να επαναλάβω και να ενισχύσω το μήνυμα που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο Ευρωπαϊκός Κώδικας ε, συμπεριφοράς ε, και κατ' ουσίαν είμαστε ευγνώμονες στην Κομισιόν που μας έδωσε τη δυνατότητα να τον συμπεριλάβουμε και εμείς ε, στο, στο διαδίκτυο. Εμείς εκπροσωπούμε 5.000 ε, ανθρώπους ε, περίπου και έχουμε αναπτύξει κάποια consensus papers όπως λέγονται είναι θεραπείες ε, για την ποιότητα ζωής και το καθεξής. Έτσι λοιπόν αυτά τα έγγραφα, γιατί έγγραφα κατ' ουσίαν είναι, υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι σε εθνικό επίπεδο ε, δεν τους αποδίδεται ιδέουσα προσοχή. Αυτό λοιπόν που κάναμε πέρυσι είναι το εξής. Ε, όπως ήδη αναφέρθηκε, ε, ξεκινήσαμε το MS βαρόμετρο, ένα είδος κριτηρίου για όλα τα κράτη-μέλη που ξεπερνάει όχι μόνο τις παρεχόμενες πλησίες αλλά και την πρόσβαση στη θεραπεία και πολλά άλλα. Και αυτό θα το επαναλαμβάνουμε κάθε χρόνο και ελπίζουμε, με την πάροδο των ετών να υπάρξει κάποια βελτίωση. Εξάλλου ζητήσαμε από τις οργανώσεις μέλη να οργανώσουν και στρογγυλές ε, τράπεζες για θέματα υγείας όπου μπορούμε να προσκαλέσουμε τον Υπουργό ε, κάποιον από τον ασφαλιστικό τομέα και βεβαίω και εκπρόσωπο των επαγγελματιών και των πασχόντων και όλοι αυτοί να συζητήσουν στο πλαίσιο της στρογγυλής τράπεζας για τα στοιχεία τα οποία ενδεχομένως μπορεί και να τους εμπνεύσουν για να επιδιώξουν κάποια αλλαγή. Αυτό το πράξαμε πέρυσι στη Σλοβενία, ε, το κάναμε και στην Ουγγαρία και για φέτος προγραμματίζουμε και άλλες τέτοιου είδους ε, στρογγυλές ε, τράπεζες. Το Κοινοβούλιο βέβαια θα μπορούσε να απευθυνθεί στο Συμβούλιο Υπουργών, στο σύνολό του και αυτό θεωρούμε ότι θα ενίσχυε περαιτέρω τις δραστηριότητές μας. Ευχαριστώ πολύ. Proszę Państwa, więc tu μας αναφέρατε διάφορα βήματα τα οποία θα μπορούσαμε να σημειώσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να συντάξω μια επιστολή που θα περιγράφει την κατάσταση στην Πολωνία και θα τη στείλω στο Πολωνικό Υπουργείο Υγείας. Αν έχετε τις στατιστικές που αναφέρατε προηγουμένως, σας παρακαλώ να μας τις δώσετε να μας αφήσετε φεύγοντας. Θα γράψω και στον Υπουργό Υγείας Καταλωνίας. Και θα του μιλήσω για την αφορά του κυρίου Ρικέλ Φελίπ. Είπατε ότι διαφορετικές περιοχές ε, προβλέπουν διαφορετική θεραπεία για τους πάσχοντες από κατά πλάκα. Αν έχετε οποιαδήποτε αποδεικτικά στοιχεία, επίσης να μας τα υποβάλλετε. Ο κύριος Στανισεύσκη, η κυρία Στανισεύσκη είπε πολύ σωστά ότι η Κομισιόν θα πρέπει να μας πει κάποια πράγματα. Ο κύριος Τατάιμ είπε ότι γίνονται έρευνες από τα κράτη-μέλη για το θέμα αυτό. Ίσως θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε προς την Κομισιόν για να συντάξει μία έκθεση για το θέμα αυτό. Φυσικά θα αφήσουμε αυτές τις αναφορές ανοιχτές, θα παρακολουθήσουμε την κατάσταση και θα δούμε τι εξελίξεις θα υπάρξουν. Ο κύριος Κάσμαν και η κυρία Στανισεύσκα και ο κύριος Σάντερ επίσης συμφωνούν, γνέφουν καταφατικά. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους αναφέροντες πάνω απ' όλα που ήρθαν να μιλήσουν εδώ. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, πολύτιμο θα έλεγα, το να έρχονται οι ίδιοι αναφέροντες στην Επιτροπή μας. Ιδίω όμως για ένα τέτοιο φορτισμένο θέμα όπως αυτό εδώ. Και τώρα περνάμε Στην αναφορά 1242 του 2007 θα δώσω το λόγο ε, στην ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τους προλαλήσαντες για να σε εκφράσω όλη μου τη συμπάθεια και όλη μου την υποστήριξη απέναντι στα άτομα που πάσχουν από την αρρώστια αυτή κατά καταπλάκας. Αυτούς που είναι εδώ σήμερα παρόντες, αλλά και τους υπόλοιπους οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην Ευρώπη. Η Ιταλική αναφορά συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τις αναφορές που μόλις συζητήσαμε. Ε, αφορά το θέμα της πρόσβασης ε, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και αφορά πιο συγκεκριμένα την ε, επιστροφή των εξόδων για τα φάρμακα και τη χρηματοδότηση των εξόδων αυτών από τις εθνικές αρχές. Πρόκειται για ένα θέμα τρομερά ευαίσθητο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι η πρόσβαση των ασθενών σε ορισμένες θεραπείες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την χρηματοδότηση των θεραπείων αυτών από τις αρχές, ειδικά όταν πρόκειται για μακροχρόνιες θεραπείες οι οποίες κοστίζουν και πολύ ακριβά. Δεν νομίζω ότι είναι χρήσιμο να επανέλθω και να επαναλάβω τα όσα υπόθηκαν ε, σε ό,τι αφορά τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό είναι πολύ λίγες. Ε, υπάρχει το άρθρο 152 που ανέφερε ο συνάδελφος της συνθήκης που λέει ότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα για την οργάνωση των συστημάτων υγείας και για την οργάνωση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αναγνωρίζουμε ότι κάθε κράτος έχει την ελευθερία να καθορίσει τον κατάλογο φαρμάκων που επιθυμεί να αποζημιώσει και τις προϋποθέσεις από τις οποίες αποσμιώνει τα έξοδα αυτά. Πρόκειται για καθαρά εθνική αρμοδιότητα, το ξαναλέω. Και ω ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο θα πρέπει να σεβαστούμε αυτήν την αρμοδιότητα. Είναι αδύνατο λοιπόν για μα, ω Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να επιβάλλουμε στι εθνικέ αρχέ το να ε, αποζημιώσουν του ασθενεί ε, για τα έξοδα που κάνουν για κάποια φάρμακα, για κάποια κατηγορία φαρμάκων. Ο ρόλο μα είναι απλώ να οργανώσουμε ένα διάλογο μεταξύ των κρατών μελών, να προαγάγουμε τις ανταλλαγές απόψεων, τόσο ώστε κάθε κράτος μέλο να γνωρίζει τι συμβαίνει στο άλλο κράτος μέλο, στο διπλανό του. Να γνωρίζει ποια φάρμακα εντάσσονται στο κατάλογο που καλύπτονται από τις αρχές και ποια όχι. Η Κομισιόν καταλαβαίνει την κατάσταση των ασθενών βέβαια, που θα ήθελαν να επιστρέφονται τα ιατρικά έξοδα ε, την απογοήτευσή του πολύ συχνά, αλλά θα ήθελα να καλέσω του πάσχοντες και τι οργανώσει του να στραφούν κυρίω και κατά προτεραιότητα προ τι εθνικέ αρχέ για να υποβάλουν αυτά τα επιχειρήματα. Τώρα έχουμε μπροστά μα μια αναφορά από έναν Ιταλό ε, υπήκο. Μόνο οι Ιταλικέ αρχέ μπορούν να επιτρέψουν την αποζημίωση στην επικράτειά του φαρμάκων που χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς ε, που πάσχουν από σκλήσει κατά πλάκα. Δεν μπορούμε έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή η συνθήκη ή οι συνθήκες γενικά να επιβάλλουμε στις Ιταλικές αρχές να ε, εντάξουν το α ή το β φάρμακο στον κατάλογο των φαρμάκων που αποζημιώνουν. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, αν δεν θέλει κανένας να πάρει το λόγο, θα ήθελα να κάνω μια πρόταση. Προτείνω να γράψουμε και εδώ μια επιστολή στο Υπουργείο Υγείας της Ιταλία αυτή τη φορά. Και πάμε στο σημείο 12. Έχουμε δύο αναφορές, την 1016 του 2007 και την 239 του 2008. Η κυρία Τερέζα Ματούλκα ίσως είναι εδώ, παρούσα, ή κάποιος άλλος ο οποίος θα την εκπροσωπήσει. Μπορεί κάποιος, η κυρία Ματούλκα, ε, να μιλήσει. Όχι. Θα δώσω το ξανά το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι δύο αναφορές αυτές είναι ουσιαστικά της ίδιας με τις προηγούμενες. Βέβαια, αφορούν την αποζημίωση φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία ε, των σπάνιων ασθενειών ε, που αντιμετωπίζονται με τα λεγόμενα ορφανά φάρμακα. Το θέμα των φαρμάκων είναι δύσκολο θέμα, αμφίσιμο σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι ένα θέμα το οποίο δυσκολεύει ακόμη περισσότερο στην περίπτωση που τα φάρμακα είναι ορφανά φάρμακα, τα οποία είναι εξαιρετικά ακριβά, αλλά είναι και απαραίτητα για τα άτομα που πάσχουν από αυτές τις σπάνιες αρρώστιες. Και εδώ η αρμοδιότητα είναι δυστυχώ εθνική και αυτό εξηγεί ότι η ίδια θεραπεία μπορεί στο α κράτος μέλος να ε, καταβάλλεται να πληρώνεται από τις εθνικές αρχές, να καλύπτεται δηλαδή από το, το σύστημά τους, αλλά σε ένα άλλο κράτος όχι. Και εδώ πάλι το, σε νομικό επίπεδο δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του ε, προτεραιότητες προϋπολογισμού σε ό,τι αφορά την επιστροφή των εξών των φαρμάκων και τις δικές του προτεραιότητες ό,τι αφορά τη δημόσια υγεία. Ε, κάνω έκκληση στους ασθενείς και στις οργανώσεις τους να στραφούν κατά προτεραιότητα προς τις εθνικές αρχές για να εκφράσουν τα επιχειρήματά τους και να προσπαθήσουν να βρουν ικανοποιητικές απαντήσεις στις διεκδικήσεις τους. Ε, τονίζω ακόμα μια φορά, είναι θεμητότατες αυτές οι διεκδικήσεις για ανθρώπους που έχουν ανάγκη από μακροχρόνιες, δύσκολες ε, θεραπείες και δαπανηρές προφανώς.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 Czy ktoś chciał zabrać θέλει να πάρει το λόγο για αυτό το θέμα. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα προς την Κομισιόν. Σε ορισμένες χώρες αυτά τα φάρμακα είναι πιο φθηνά ε, από ό,τι στην Πολωνία. Παραδείγματος χάρη στη Γερμανία είναι πιο φθηνά αυτά τα φάρμακα. Διερωτώ με, δεν θα μπορούσαν οι ασθενείς να αγοράσουν τα φάρμακα αυτά όπου είναι φθηνότερα και όχι να τα αγοράσουν στη χώρα που ζούνε. Oui, Monsieur le Président, je, vous remercie pour, euh, pour... Κομισιόν, ευχαριστώ πολύ για το ερώτημά σας, Πρόεδρε. Υπάρχει η ελεύθερη κυκλοφορία και των προσώπων και των αγαθών. Είναι δύο από τις βασικές ελευθερίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι απόλυτα δυνατό να εισαχθεί από το εξωτερικό το τάδι το δίνα φάρμακο και μπορούν και οι ασθενείς να υποστούν θεραπεία σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα της πρόσβασης στη, στο υγειονομικό σύστημα άλλων χωρών το θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των ασθενών είναι ε, αντικείμενο ε, πρότασης Κομισιόν που συζητείται αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, σκοπό έχουμε να διευκολύνουμε στο μέλλον την ε, παροχή υπηρεσιών υγειονομικής ε, φύσεως και φαρμάκων σε ασθενείς που θα ήθελαν να υποφεληθούν από τέτοιες θεραπείες και φάρμακα στο εξωτερικό. Πρόεδρος. Πολύ ωραία. Θα ενημερώσουμε τους αναφέροντες για τα όσα μας είπε η Κομισιόν. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτές τις αναφορές. Μόνο και μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους. Θα κρατήσουμε ανοιχτές αυτές τις αναφορές και δεν θα, τους, δεν θα κλείσουμε αυτό το παραθυράκι που έχουν ε, οι αναφέροντες. Πάμε στο σημείο 13, στην αναφορά 1012 του 2007 και στην αναφορά 1234 του 2007. Ο Χουάν Μαρία Μαρτίνες Φερνάντες είναι εδώ στην αίθουσα, παρακαλώ. Ή κάποιος εκ μέρους του αναφέροντος, ο κύριος Φερέρο. Ναι, είναι εδώ. Κύριε Φερέρο. Καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Ε, αξιότιμοι κύριε, εξ ονόματος της ε, ε, Ένωσης των Εργαζόμενων στην Ισπανία, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την προσοχή σας έναντι αυτής της αναφοράς που υποβάλαμε και που θεωρούμε ότι είναι δικαιολογημένη όσον αφορά το πνεύμα αλλά και το γράμμα της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ουχετέ ε, προσπαθεί να προωθήσει τα συναδεξιοδοτικά συστήματα για τους εργαζόμενους και ε, προσανατολιζόμαστε βεβαίω στα πλεονεκτήματα των εργαζόμενων. Ε, σήμερα δεν θα παρουσιάσουμε πάλι το περιεχόμενο της δικής μας αναφοράς, αλλά θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε εκείνες τις πτυχές που θεωρούμε ότι έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Ο στόχος της οδηγίας 80 987 είναι η προστασία των εργαζόμενων στην περίπτωση αφαιρεγγιότητας της επιχείρησης. Το άρθρο 8 αυτής της οδηγίας αναφέρεται ειδικά στα δικαιώματα των εργαζόμενων όσον αφορά τις συμπληρωματικές συντάξεις στην περίπτωση αφαιρεγγιότητας της επιχείρησης. Η μεταφορά στο ισπανικό δίκαιο αυτής της οδηγίας ε, συμπίπτει με την ε, εξωτερήκευση ή με τη δημιουργία κάποιων εξωτερικών ε, ταμείων που θα έχουν σαν αποστολή να καλύπτουν τις συνταξιοδοτικές υποχρεώσεις μιας επιχείρησης σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας. Και αυτό οδηγεί σε μια μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα όσον αφορά την κατοχήρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτή η εξωτερήκευση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων έχει δεσμευτικό χαρακτήρα για όλες τις επιχειρήσεις και για όλους τους οικονομικούς τομείς. Ωστόσο ταυτόχρονα υπάρχει μια μεταβατική διάταξη βάσει της οποίας ο ιδιωτικός τομέας, οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές εταιρείες μπορούν να διατηρούν τις συνταξιδοτικές υποχρεώσεις έναντι των εργαζομένων υπό τη μορφή εσωτερικών ε, ταμείων. Αυτή η διακριτική μεταχείριση συνεπάγεται μία διάκριση ε, για όλες τις ε, επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν σε αυτή τη μεταβατική διάταξη γιατί ακριβώς ζημιώνονται τα δικαιώματα των εργαζόμενων του χρηματοοικονομικού τομέα. Και αυτό για τρεις λόγους. Γιατί όσον αφορά τη βιωσιμότητα των συντάξεων σε περίπτωση εμφαρικιότητας της επιχείρησης, σε μια κατάσταση μεγάλης ανασφάλειας οι ισπανικές αρχές επανέλαβαν για να υπερασπιστούν αυτή τη διακριτική μεταχείριση για τον χρηματοπιστωτικό τομέα την ε, αξιοπιστία των ισπανικών χρηματοπιστωτικών οργανισμών και τους αυστηρούς ελέγχους των οικονομικών αρχών. Παρακάμπτοντας τις ε, περιπτώσεις εκείνες ε, αφαιρεγγιότητας. Μόνο στη δεκαετία του 80 ε, υπήρξαν ε, δέκα χιλιάδες εκατομμύρια ευρώ ε, για τις συμπληρωματικές συντάξεις των εργαζόμενων στην τράπεζα Σανταντέρ, τα οποία όμως δεν δόθηκαν στους εργαζόμενους. σε περιπτώσεις χρεοκοπίας ε, αυτό είναι κατάφορα σε βάρος των εργαζόμενων. Όσον αφορά την εξωτερήκευση αυτών των συνταξιδοτικών ε, ταμείων και αυτή η εξέρεξη που υπάρχει για το χρηματοπιστωτικό τομέα δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση στην Ισπανία. Η τράπεζα του Σανταντέρ έχει εσωτερικά ταμεία για τις συμπληρωματικές συντάξεις των εργαζόμενων που ανέρχονται πάνω σε 10.000 εκατομμύρια ευρώ. Αυτή η έλλειψη ασφάλειας οδήγησε το συνδικάτο μας να απευθυνθεί προς την Τράπεζα της Ισπανίας γιατί οι πρικοδοτήσεις στα, στο ιστορικό ταμείο συνταξιοδοτήσεων ήταν ανεπαρκής. Και Η οδηγία 80, 987 αναφέρεται στην προστασία όχι μόνο σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας των κεκτημένων δικαιωμάτων, αλλά αναφέρεται και στις συμπληρωματικές παροχές η βασική διαφορά μεταξύ των εσωτερικών ταμείων και εξωτερικών ταμείων είναι η εξή. Τα εσωτερικά ταμεία είναι η ιδιοκτησία της επιχείρησης, συνεπώς είναι ένα εργαλείο ρευστότητας της επιχείρησης, ενώ τα εξωτερικά ταμεία είναι ιδιοκτησία των εργαζόμενων και συνεπώς είναι εγγυημένα ε, μέσω οργανισμών που είναι εξωτερικοί προς την επιχείρηση. Όπως είναι προφανές, ε, τα δικαιώματα των εργαζόμενων ε, στην επιχείρηση ε, κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου είναι καθοριστικά στοιχεία. Αυτή η κατάσταση αττική στη διάκριση των εργαζόμενων στη τράπεζα Σανταντέρ σε σύγκριση με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της ε, εξαίρεσης της Τράπεζας Σανταντέρ από την ε, διάταξη αυτή. Με τον τρόπο αυτό, οι εργαζόμενοι της τράπεζας αυτής υφίστανται διακριτική μεταχείριση όσον αφορά την ελεύθερη διακίνηση μέσω των, ε, προς τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παραμονή στην επιχείρηση ο όρος μάλλον παραμονή στην ε, επιχείρησή τους ε, δυσχεραίνει την κινητικότητα των εργαζόμενων αυτών ε, είτε προς μια άλλη Ισπανική τράπεζα, είτε προς μια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Γιατί εφόσον μετακινηθεί ο εργαζόμενος θα χάσει τις συμπληρωματικές συντάξεις, δικαιώματα τα οποία παραμένουν στην κατοχή των επιχειρηματιών και δεν μεταφέρονται κατά κανένα τρόπο στους ίδιους τους εργαζόμενους. Δεν υπάρχει λοιπόν η συμμεταχείριση όσον αφορά τη διατήρηξη του δικαιώματο συνταξιοδότη, γιατί η νομοθεσία μα δεν εγγυάται αυτή την ίση μεταχείριση σε περίπτωση μετακίνηση των εργαζομένων. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η εξαίρεση του χρηματοπιστωτικού τομέα βασίζεται στην ύπαρξη, όπω ήδη είπαμε, μια μεταβατική διάταξη στην Ισπανία, η οποία εισήχθη στον Ισπανικό νόμο το 1995 μέσω του νόμου για τις ιδιωτικές ασφάλειες. Πέρασαν 14 χρόνια κυρίες και κύριοι και μια μεταβατική διάταξη η οποία είχε ακριβώς ένα μεταβατικό χαρακτήρα έχει εδρεωθεί. Εμείς ε, διατυπώσαμε πάρα πολλά αιτήματα προς το Εργατικό Δικαστήριο της Ισπανίας σε σχέση με τα συνταξιοδοτικά ταμεία των εργαζόμενων στο χρηματοπιστωτικό τομέα εν γέννη και στην Τράπεζα Σανταντέρ ειδικότερα. Ε, θέσαμε στα δικαστήρια αυτά ως ε, ε, βασικό ερώτημα το οποίο ποτέ δεν απαντήθηκε ε, σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Και είπαμε ότι υπάρχει εδώ μια κατάφορη παραβίαση του άρθρου ε, της συνθήκης του Άμστερνταμ που οδηγεί την Επιτροπή στην υποχρέωση εφαρμογής του άρθρου 69. Η η οδηγία 80-987, η οδηγία 98-49 και η συνθήκη του Άμστερνταμ στο άρθρο 39, εδάφιο 3, ε, καθώς και το άρθρο 234 της ίδιας συνθήκης ε, σε σχέση με την παραπομπή στο ΔΕΚ όταν ε, τίθεται ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να λυθεί με τα εσωτερικά δικαιοδοτικά όργανα ε, όλα αυτά καταδεικνύουν ε, πόσο τεκμηρωμένο είναι το αίτημά μας. Ε, θέλουμε να πούμε ότι εδώ ότι ο, ο Ισπανός διαμεσολαβητής δύο φορές αποφάνθηκε υπέρ της εξωτερήκευσης των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων για όλους τους εργαζόμενους του χρηματοπιστωτικού ε, τομέα ε, το 2002 και το 2004. Ε, ζητούμε λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει δεκτό το αίτημά μας, την αναφορά μας και να πιέσει την Ισπανική κυβέρνηση να καταργήσει τη μεταβατική διάταξη ε, του νόμου για τις ιδιωτικές ασφάλειες που ακριβώς παρεμποδίζει τις, ε, την κινητικότητα των εργαζόμενων. Thank you Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να πω ότι η Κομισιόν έχει απόλυτη κατανόηση Απόλυτη κατανόηση λοιπόν για το θέμα που είναι πολύ περίπλοκο και θα ήθελα να προσπαθήσω να το εξηγήσω όσο πιο εύκολα μπορώ. Η συγκεκριμένη ισπανική νομοθεσία Όσον αφορά τις επικουρικές ε, συντάξεις διαχωρίζει μεταξύ του, συνόλου της οικονομίας και συγκεκριμένων τομέων. Έχουμε με βάση την Ισπανική νομοθεσία κάποια ειδικά ταμεία που εγγυώνται ότι ο εργαζόμενος ε, που μετά από κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο δεν εργάζεται πλέον καταβάλει, συνεχίζει να καταβάλει τις εισφορές του. Στον ε, χρηματοπιστωτικό τομέα ε, υπάρχει διαφάνεια. Οι χρηματοψηφιακοί οργανισμοί δεν επιτρέπουν να το κάνουν αυτό. Δημιουργούν δικά τους εσωτερικά αποθέματα και σε περίπτωση πρόορης συνταξιοδότησης τότε ε, ο τομέας ενδέχεται και ο ενδιαφερόμενος ενδέχεται να απολέσει τα συνταξιωτικά του δικαιώματα. Αυτή η κατάσταση υπάρχει και σε άλλα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν έκρινε ότι είναι απαραίτητο το θέμα να εξεταστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η Κομισιόν ανέλησε λοιπόν την κατάσταση και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να θεσπιστεί οδηγία η οποία θα διευκρινίζει ε, τα δικαιώματα των εργαζομένων σε τέτοιου είδου περιπτώσει, γιατί ενδεχομένω να γνωρίζετε ότι και το Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Η Κομισιόν κατέθεσε μια οδηγία για τη δυνατότητα μεταφορά συνταξιδοτικών δικαιωμάτων εργαζομένων. Ε, τώρα το όλο θέμα έχει κατευθύνει στο Συμβούλιο για πρώτη ανάγνωση και μετά θα προχωρήσει. Θα επανέλθω αργότερα να σα εξηγήσω γιατί η κατάσταση είναι τόσο περίπλοκη. Η οδηγία λοιπόν αυτή αυτή βασίζεται στα άρθρα 39 και 42 της ε, ε, οδηγίας περί της ελεύθερης μετακίνησης των εργαζομένων και εξετάζεται μια κατάσταση όπου ας πούμε ένας Ισπανός εργαζόμενος σε τράπεζα φεύγει από αυτή την Ισπανική τράπεζα και πάει σε μια άλλη χώρα. Τότε η οδηγία είναι σαφής για τα συνταξιωτικά δικαιώματα του εν λόγω ανθρώπου. Η Κομισιόν όμως θεώρησε ότι είναι δύσκολο να ε, διαφοροποιήσει κανείς την κατάσταση αυτή από μια άλλη περίπτωση όπου ένας εργαζόμενος φεύγει από μια συγκεκριμένη Ισπανική τράπεζα και πάει να εργαστεί κάπου αλλού. Γι' αυτό λοιπόν την πρόταση οδηγίας δεν τη στήριξε μόνο στο 39 και το 42 της συνθήκης αλλά και στο άρθρο 94 της συνθήκης. Γιατί με τον τρόπο αυτό θα ε, λύνονται, θα ρυθμίζονται καταστάσεις που δεν αφορούν διασυνοριακή εργασία. Ε, κρίθηκε λοιπόν να χρησιμοποιηθεί και το συγκεκριμένο άρθρο της ε, εσωτερικής αγοράς έτσι ώστε να καλύπτεται η δυνατότητα μετακίνησης και μέσα στην επικράτεια μιας και μόνο χώρας. Βέβαια αυτή η οδηγία δεν έχει ακόμα τεθεί σε ισχύ, ε, τώρα είναι προς εξέταση στο Συμβούλιο μετά από τη θετική γνωμοδότηση του Κοινοβουλίου, άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε αυτή την οδηγία. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να εφαρμόσουμε τη συνθήκη και θα ήθελα να σχολιάσω το άρθρο 39 που αφορά στην ελεύθερη μετακίνηση ατόμων και αν δει κανεί τον τρόπο με τον οποίο το 10 αντιμετώπισε αυτό το άρθρο θα διαπιστώσει ότι το ΔΕΚ είπε ότι όταν υπάρχει ξεκάθαρη διακριτική μεταχείριση πρέπει να υπάρχει και παρέμβαση. Διακριτική μεταχείριση αυτό αφορά ανθρώπους με ε, διαφορετική ηθαγένεια αλλά και διαφορετική μεταχείριση σε άνθρωπα τα οποία μετακινούνται στην επικράτεια μιας και μόνο χώρας και σε άλλα που ε, μετακινούνται εκτός της χώρας. Η ισπανική τώρα περίπτωση δεν αφορά κάποιον που έτυχε διαφορετική μεταχείριση επειδή έφυγε από την Ισπανία. Η ισπανική περίπτωση είναι ότι ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ε, έτυχε διαφορετική μεταχείριση, έτυχε και να είναι στο χρηματοψηφιακό τομέα αντί να εργάζεται σε κάποιο άλλο τομέα. Σύντομα λοιπόν, η άποψη των νομικών υπηρεσιών της Κομισιόν είναι ότι η άμεση παραβίαση του άρθρου 39 ισχύει μόνο σε καθαρά υποθετικές περιπτώσεις. Δηλαδή αν υποθέσουμε ότι κάποιος από το χρηματοψηφικό τομέα δεν πάει σε εταιρεία άλλης χώρας λόγω της έλλειψης διατάξεων δεν μπορεί να τεκμηριωθεί και η όλη υπόθεση. Αυτό είναι βέβαια καθαρά υποθετικό. Τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά αν είχαμε συγκεκριμένη περίπτωση Ισπανού από τον τραπεζικό τομέα που να μπορεί να αποδείξει ότι δεν μπορεί να δεχθεί εργασία σε άλλη χώρα λόγω του κινδύνου απώλειας των ε, συνταξιδοτικών του δικαιωμάτων ή όπου ε, κάποιος να μπορεί να ισχυριστεί ότι ε, έφυγα και έχασα τα ε, στεξιωτικά μου δικαιώματα. Αυτό δεν θα ήταν υποθετική περίπτωση. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι για να τεκμηριωθεί παραβίαση χρειαζόμαστε και άλλα στοιχεία πέρα από απλές παραδοχές. Όμως η πολιτική της Κομισιόν είναι να λάβουμε αυτή την υπόθεση πολύ σοβαρά γιατί ενδέχεται η περίπτωση αυτή να εμφανιστεί και σε άλλες χώρες. Ε, και γι' αυτό τον λόγο έχουμε δρομολογήσει και αυτή την περίφημη οδηγία ε, περί ε, μετακίνησης εργαζομένων το θέμα της οδηγίας περί αφαιρεγγιότητας είναι διαφορετικό και αυτό θα σας το αναλύσει ο συνάδελφός μου. Πρόεδρος, θα ήθελα μόνο να σας ε, παρακαλέσω να εκφράζεστε σύντομα γιατί ε, δυστυχώς έχουμε, μας υποποιήσει χρόνο και αν έχετε καλοσύνη να καταλήξετε και κάπου. Κοιτάξτε, αυτή η οδηγία περί αφαιρεγγιότητας προβλέπει τη δυνατότητα επικουρικής, καταβολής επικουρικής σύνταξης σε περίπτωση ε, ε, του εργοδότη. Αλλά εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν ποια μέτρα πρέπει να λάβουν. Δεν ε, υπάρχει καμία συγκεκριμένη οδηγία, ε, δεν έχει προτείνεται κανένα συγκεκριμένο μέτρο σε αυτό το άρθρο. Γι' αυτό λοιπόν και τα κράτη-μέλη ενέκριναν διαφορετικά μέτρα για να εφαρμόσουν το άρθρο αυτό. Μόλις πρόσφατα η Κομισιόν τον Απρίλιο του περασμένου έτους ε, σύστη στα κράτη-μέλη να συμμορφωθούν με το άρθρο αυτό. Και όσον αφορά στον τραπεζικό τομέα της Ισπανίας, η Κομισιόν διαπίστωσε ότι το να υπάρχει πρόβλεψη για τη διατήρηση εσωτερικών ταμείων, αυτό επιτρέπεται με βάση συγκεκριμένα μέτρα που έχουν σχέση με διοικητική, διοικητικό έλεγχο που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον εξίσου αυστηρός όπως και τα εξωτερικά εργαλεία. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν πιστεύει ότι το άρθρο αυτό επιτρέπει τη λήψη τέτοιων μέτρων. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα ήθελα τώρα να ρωτήσω ποιος επιθυμεί να λάβει το λόγο. Ελασέντερ, Σάντσες και νομίζω ότι κατόπιν κλείνει ο ε, κατάλογος των μιλητών. Ε, η κυρία Ελασέντερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι αναγνωρίζοντας δικαιολογημένα ότι η Ισπανική κυβέρνηση σε αυτή την περίπτωση κρίσης προσπαθεί να έχει ένα μεγαλύτερο έλεγχο. Από την άλλη είναι αλήθεια ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία της απάντησης της Κομισιόν που με κάνουν να προβληματιστώ. Και θα ήθελα να μου τα η Επιτροπή. Το άρθρο 8 της οδηγίας ε, προβλέπει ότι θα πρέπει, ε, μπορούν ε, να έχουν εσωτερικά ταμεία οι επιχειρήσεις. Αλλά αυτό αναφέρεται ως ε, μεταβατική διάταξη. Και θα ήθελα να ρωτήσω πού έγκυται η μεταβατικό, το μεταβατικός χαρακτήρας αυτής της διάταξης. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα μιας μεταβατικής διάταξης. Επίσης λέγεται ότι θα πρέπει να υπάρχει αυστηρός έλεγχος σε αυτά τα εσωτερικά ταμεία. Ε, να δούμε κατά πόσο πληρούνται κάποιε εξίσου αυστηρέ προποθέσει στα εσωτερικά ταμεία όπως ισχύει και με τα εξωτερικά ταμεία επικουρικών συντάξεων. Ε, όσον αφορά μια νέα οδηγία για την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων περιπτώσεων ε, που οδηγούν σε μια που οδηγούν σε μια υπονόμευση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Θα ήθελα να ρωτήσω, ε, στην περίπτωση που θα εγκριθεί μια τέτοια οδηγία, η παρούσα κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή ε, θα βελτιωθεί. Για παράδειγμα, αν η οδηγία αυτή την οποία συζητούμε και αναγνωρίζει ότι εδώ είναι κάπως ευάλωτα τα δικαιώματα των εργαζόμενων όσον αφορά την κινητικότητά τους. Ε, Προφθέτει ότι όταν εγκριθεί η οδηγία αυτή από την Κομισιόν μετά την πρώτη ανάγνωση, αυτό σημαίνει θα μπορούν τα συνδικάτα να υποβάλουν κάποια αιτήματα, να πετήσουν τα δικαιώματά τους σε σχέση με την οδηγία αυτή. Ο κύριος Σάντσεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να τονίσω την ε, σημασία αυτής της συζήτησης γιατί ε, πραγματικά ε, δεν θα πρέπει να θέσουμε σε κίνδυνο τα συνταξιδοτικά ταμεία και θα πρέπει οι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερες εγγυήσει για τα δικαιώματά τους και να διευκολυνθεί η κινητικότητά του. Αυτά τα αιτήματα είναι και τα δύο απολύτω θεμητά. Τώρα, όσον αφορά τα ερωτήματα που διτύπωσε προλύσασα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Υπάρχει ένα θέμα, εσωτερικό ταμείο, εξωτερικό ταμείο. Είναι προφανές ότι η οδηγία εξετάζει και τις δύο δυνατότητες και στο χρηματοπιστωτικό κλάδο ενδεχομένως μπορεί να μην είναι υποχρεωτικό ένα εξωτερικό ταμείο. Οι εγγύησεις εδώ διαφέρουν από ό,τι για τις λοιπές επιχειρήσεις και υπάρχονται σε πιο αυστηρές απαιτήσει από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Συνεπώς θα πρέπει να μας πει η Κομισιόν πώς ε, βλέπει τον μεταβατικό χαρακτήρα αυτού του ταμείου. Το άλλο αφορά την εδραίωση και το χείρο των δικαιωμάτων των εργαζομένων τα επικουρικά δικαιώματα είναι δυνητικά δικαιώματα, ενδυνάμει δικαιώματα. Για να προσεγγίσουμε αυτό το θέμα υπάρχουν δύο τρόποι. Το πρώτο είναι οι συλλογικέ διαπραγματεύσει. Είναι πολύ σημαντικό να, γίνουν, να προχωρήσουν σε όλα τα επίπεδα οι συλλογικέ διαπραγματεύσει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και το άλλο θέμα αφορά τα, την νομοθεσία της ε, κοινότητας που θα πρέπει να διευκολύνει την κινητικότητα των εργαζόμενων. Τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη ανάγνωση. Το Συμβούλιο ε, συναντάει πάρα πολλές ε, δυσκολίες και θα είναι δύσκολο να προσεγγιστούν όλα τα θέματα στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας ή να επιληθούν τα θέματα ε, στο πλαίσιο αυτής της οδηγίας. ή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσπαθήσει να εξεύρει άλλους ε, τρόπους επίλυσης, γιατί πρόκειται για μια συζήτηση εξαιρετικά σημαντική. Να θέσω ένα ερώτημα προς τους αναφέροντες. Θα θέλετε να αντιδράσατε στα λεγόμενα της Κομισιόν και στα ερωτήματα που έθεσαν τα μέλη της Επιτροπής μας, οι βουλευτές. Εγώ θα πρότεινα να αφήσουμε αυτή την αναφορά ανοιχτή, περιμένοντας ε, περαιτέρω πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμως, αν θέλετε να αντιδράσετε, θα σας ξαναδώσω το λόγο. Θα σας δώσω δύο ή τρία λεφτά στους αναφέροντες για να δευτερολογήσετε. Ε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα δούμε τι γίνεται. Υπάρχει μια σειρά θεμάτων. τα οποία δεν εμπόδισαν ούτε την αφαιρεγγιότητα ούτε τους, ε, την διεξαγωγή σωστών ελέγχων για τις τράπεζες. Είναι ε, Πέρα από όλα τα επιχειρήματα που προβλήθηκαν εδώ, ε, θα πρέπει να πούμε ότι το σύστημα έχει κάποια κενά. Και αυτά τα κενά ε, συναρτώνται ακριβώς με τις ε, πολυάριθμες προσφυγές στα δικαστήρια. Το ανώτατο Ισπανικό Δικαστήριο, το οποίο είναι το ανώτατο δικαιοδοτικό όργανο της χώρας, μέσω του άρθρου 234 ε, κρίνει τα θέματα αυτά. Ε, αλλά θεωρώ ότι πραγματικά εδώ διαπιστώνεται μια απώλεια των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Εάν ε, χάσουν το δικαίωμα συμπληρωματικής σύνταξης, Γιατί για να μπορεί ένας εργαζόμενος της ε, τράπεζας Santander να, αν θέλει να πάει σε μια άλλη χώρα για να εργαστεί εκεί, ε, θα χάσει τα δικαιώματά του της επικουρικής σύνταξης. Πρόκειται για μια διάκριση έναντι των εργαζομένων. Γι' αυτό ε, θεωρούμε ότι υπάρχει εσφαλμένη μεταφορά στο Ισπανικό Δίκαιο αυτής της οδηγίας γιατί υπάρχουν βεβαίως εγγυητικά ταμεία τα οποία εγγυώνται όχι μόνο στους καταθέτες αλλά και στα χρήματα και στις, τις εισφορές των εργαζόμενων ε, στην ε, τράπεζα που θα έπρεπε να συνιστούν περιουσιακά στοιχεία των εργαζόμενων. Γιατί στην περίπτωση αφαιρεγγιότητας τα περισσοκά αυτά στοιχεία χάνονται για τους εργαζόμενους. Σε περίπτωση αφαιρεγγιότητας σε μια σοβαρή οικονομική κρίση όπως αυτή που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν, δεν υπάρχει τρόπος να καταγραφεί η, η απώλεια των δικαιωμάτων των εργαζόμενων σε περιουσιακά στοιχεία όσον αφορά τα ταμεία αυτά. Πολύ θα κάνουμε αυτό που σας είπα. Θα, περιμένουμε... θα κάνουμε αυτό που είπα. Θα περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες από την Κομισιόν. Θα αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά και θα συνημερώσουμε για τις εξελίξεις. Θα ξανασυζητήσουμε αυτές τις αναφορές και θα σας προσκαλέσουμε στη συνεδρίασή μας για να παραστείτε και να αντιδράσετε. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Περνάμε στο σημείο 14 της μερικής διάταξης, που είναι η έκθεση Μαγκίνες. Ναι. Κύριε Μαγκίνε, έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, από αυτή τη γωνία δεν μπορώ να, να σας δω κατάματα. Κοιτάξτε, ναι, τώρα κοιτάω και σας βλέπω. Ζητώ συγγνώμη προ όλου, γιατί βγαίνω συνέχεια, αλλά έπρεπε να βοηθήσω κάποιο, κάποια ομάδα <clears throat> επισκεπτών. Θα είμαι σύντομη γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Η έκθεση αυτή ε, έρχεται εδώ για να χρωματίσει την ε, ζωή μας. Ε, συνήθως η ζωή μας είναι σε μαύρο και άσπρο. Ε, τώρα όμως έχουμε μια χρωματιστή έκθεση ε, χάρη στις στατιστικές της δουλειάς της Επιτροπής Αναφορών τα περισσότερα χρόνια. Αυτό το καταφέραμε χάρη στη βοήθεια της Γραμματείας. Μπορείτε να δείτε ποιες είναι οι αναφορές, από ποιες χώρες έρχονται, τι τομείς αφορούν κτλ. Πέρα από τις ευχαριστίες προς τη Γραμματεία για τη βοήθεια που μου προσέφερα, θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Κομισιόν που από την αρχή πραγματικά μου έδωσε πολύτιμη βοήθεια στη σύνταξη της έκθεσης. Δύο-τρία λόγια θέλω να σας πω. Για να εργαστούμε καλύτερα εμείς, πρέπει οι πολίτες να καταλάβουν τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, γιατί εξουσία έχουμε για να το κάνουμε. Και νομίζω ότι Κάθε χρονιά θα πρέπει να είμαστε καλύτεροι από την προηγούμενη. Αυτό το αναφέρω στην έκθεση. Η Ιρλανδία, Φερρυπίν, έχει το μεγαλύτερο αριθμό αναφορών κατά κεφαλήν σε σχέση με τα άλλα κρατημέλη. Ίσως επειδή έχουμε πολλούς Ιρλανδούς σε αυτή την επιτροπή. Και επομένως οι Ιρλανδοί έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της δουλειάς της ε, Επιτροπής Αναφορών. Ανέφερα τις στατιστικές, ε, ίσως ε, θα σας βοηθήσουν, θα μπορούσατε να τις σχολιάσετε αν θέλετε. Γίνεται λόγος για ό,τι κάνουμε πέρυσι. Ε, την προσοχή στο πώς συνδεόμαστε με τους πολίτες ε, για τη δουλειά που κάνουμε. Ορισμένοι μας σαν το φτωχό συγγενή. Κι όμω είμαστε η Επιτροπή που έχουμε τη μεγαλύτερη άμεση επαφή με του Ευρωπαίου πολίτε. οι οποίοι έρχονται εδώ πέρα για θέματα που του απασχολούν, ε, για θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τι φαματερές, τι συντάξει του. Είμαστε σημαντική Επιτροπή. Και αν περάσει από όλα τα μέλη η, συνθήκη της Λισαβόνας, ε, νομίζω θα ενισχυθεί το έργο μας. Ε, αναγνωρίζουμε τη βοήθεια του διαμεσολαβητή, ήταν εδώ σήμερα πριν από λίγο και τη σημασία των αποστολών ε, για την εξέβρεση στοιχείων και την ε, ε, συγγραφή κάποιων πορισμάτων. Είχαμε πάρα πολύ σημαντικά θέματα, πολιτικά ευαίσθητα, όπως η έκθεση για, τις, για το Misleading Directories, για τον αγωγό φυσικού αερίου Nord Stream. σημαντικά θέματα, τα οποία τα αναφέρει η έκθεσή μου. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι το περιβάλλον αφορούν πολλές οι αναφορές. Ίσως γιατί έχουμε πολλά νομοθετήματα σε αυτόν τον τομέα. Αυτό σχετίζεται και με ένα άλλο ερώτημα, πιο ευρύ, που δεν το εξετάζει η έκθεση αυτή, γιατί δεν είναι θέμα της έκθεσης. Έρχομαι αυτή τη στιγμή από μία συνεδρίαση με επιστήμονες, οι, οι δήμονες σε θέματα αγροτικά κτλ. Οι οποίοι μίλησαν για κάποια, κάποια διάσταση που υπάρχει ανάμεσα στο, στα θέματα των οδηγιών και κανονισμών ας και, στο, και στη γνώση των Ευρωπαίων πολιτών. Επίσης το θέμα της εφαρμογής. Εμείς έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε εδώ, όχι το ρόλο του αστυνομικού, αλλά πρέπει να δούμε τι συμβαίνει σε κάθε κρατός μέλος και να υποδείξουμε τι βελτιώσεις πρέπει να σημειωθούν. Αυτά, Πρόεδρε, λόγω ελλείψεως χρόνου. Ε, ευχαριστώ. Κυρία Μαγκίνες. Κοίταξα έτσι πολύ σύντομα την έκθεση. Είναι θαυμάσια, είναι διαφανής, είναι εύληπτη. Και δίνει, χύνει έτσι ένα νέο φως χρωματιστό φως στη δουλειά που κάνουμε σε αυτήν την Επιτροπή. Ο κ. Μαυρομάτης, ο κ. Σάτκης και ένα άλλο ομιλητή. Δύο λεπτά ο καθένα παρακαλώ. Έχουμε ακόμα μία αναφορά, παρουσία του αναφέροντος. Ο κ. Μαυρομάτης, δύο λεπτά παρακαλώ. Θα είμαι πολύ πιο σύντομος. Ε, η πολυχρωμία της έκθεσης της συναδέλφου Μαγκίνας είναι εκπληκτική αλλά είναι και ουσιαστική γιατί καταγράφονται πέραν από τα νούμερα και τους αριθμούς και τα ποσοστά όλες αυτές οι διαδικασίες που ήταν απαραίτητες για να γνωρίσουμε το πραγματικό έργο και του διαμεσολαβητή αλλά και της δικής μας Επιτροπής. Και αυτό η αγαπητή Μαγκίνες ε, το φέρνει ανάγλυφα σε εμάς ώστε να βρούμε σε αυτήν την έκθεση που σύντομα εδώ είδα μερικά από τα στοιχεία, παραδείγματα πολύ ουσιαστικά. Εκείνο το οποίο πρέπει να καταγραφεί κύριε Πρόεδρε, ότι βρίσκεται μάλιστα η έκθεση αυτή στο σύγχρονο περιβάλλον, γιατί το περιβάλλον είναι που απασχολεί παγκόσμια πλέον όλα τα κράτη και όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και βλέπω λοιπόν ότι πολλές από τις αναφορές, 309 περίπου, αφορούν το περιβάλλον. Στη συνέχεια τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό δείχνει την δική μας ευαισθησία. Η ευαισθησία δηλαδή της Επιτροπής αλλά και των αναφερόντων που φτάνουν μέχρι την δική μας Επιτροπή. Εκείνο που με, α, κυρίως όμως με ανησυχεί κύριε Πρόεδρε είναι ότι ενώ υπάρχουν βελτιώσεις σε πάρα πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αναφορές ή Υπάρχουν τα καινούργια κράτη όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία η οποία αναφέρονται πλέον και πάνε να ε, καταρρύψουν ρεκόρ προηγούμενα αναφορών κάτι που σημαίνει ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή και σε αυτό το σημείο. Η Επιτροπή μας και η συνάδελφος που επεξεργάζεται και το τελικό κείμενο. Εμείς θα έχουμε την δυνατότητα με τροπολογίες να αναφερθούμε σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι έχει κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά και εύχομαι να είναι επικοδομητική για όλη την Επιτροπή και για όλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίτσελ τώρα για δύο λεπτά επίσης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο για αυτή την έκθεση. Είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα θέματα. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικές οι επισκέψεις που κάνουμε στο εξωτερικό. Τρίτον, αν θέλουμε να είμαστε αξιόπιστοι ως ε, Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και εφόσον το Κοινοβούλιο έχει περισσότερες αρμοδιότητες μετά από την Λισαβόνα και έχουμε περισσότερες αρμοδιότητες συναπόφασης, θα έπρεπε να εξασφαλίσουμε ότι δεν δίνουμε φρούδες ελπίδες στους αναφέροντες. Δεν κάνουμε έτσι, εσωτερική δεν κάνουμε διαφήμιση για εσωτερική κατανάλωση, να ενθαρρύνουμε ας πούμε, τους ανθρώπους να έρχονται εδώ. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να εκφράζουμε αυτή τη ρεαλιστική προοπτική και προς τους ε, αναφέροντες. Δεν θα πρέπει να φέρνουμε αδίκο στον κόσμο εδώ. Ε, χάνουμε χρόνο, χάνουμε χρήμα, ξοδεύουν και εκείνοι χρόνο και χρήμα και δεν είναι καλό για το ρόλο του Κοινοβουλίου. Το μόνο που θέλω να πω είναι. Αυτά και μετά από αυτό δεν έχω να πω τίποτα άλλο πέραν του να συγχαρώ τη συνάδελφο Μαγκίνε. Ο κύριο Άτκιν, επίση δύο λεπτά. εγώ ποτέ δεν χρειάστηκε να μιλήσω δύο ολόκληρα λεπτά, λέει ο κύριο Άτκινς. Κοιτάξτε, αυτή η έκθεση είναι μια δικλίδα ασφαλεία και πρέπει ε, να επιτρέπουμε στους πολίτες ε, να εκφράζουν την απογοητευσή του. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μία F και G στα αγγλικά είναι πολύ σημαντικά. Το λέμε αυτό κάθε χρόνο. Ε, νομίζω ότι ορισμένα κράτη-μέλη πρέπει να παρακινηθούν για να είμαστε σίγουροι ότι θα απαντήσουν ε, οποτεδήποτε κληθούν. Κατόπιν εκεί που γίνεται λόγο για το προσωπικό και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Αναφέρεται πιο κάτω στο τι νομίζω και εντυπωσιάζομαι, ομολογώ, για αυτά που αναφέρονται σχετικά με την Equitable Life, την εταιρεία ε, οι συνάλφοι στη Βρετανία προσπάθησαν να κάνουν ό,τι μπορούν, αλλά το θέμα είναι ότι δυστυχώ ακόμα δεν έχει δοθεί απάντηση. Το σημαντικότερο όλων είναι η παράγραφο 9. Οι αναφέροντε δεν έχουν βέβαια πάντα δίκιο, αλλά πρέπει τουλάχιστον να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά του ε, και εμεί να την ακούσουμε. Πραγματικά είναι μια θαυμάσια, ε, έγχρωμη, χρωματιστή έκθεση και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Μαγκίνε που την συνέταξε. Δεν νομίζω κύριε Πρόεδρε ότι χρησιμοποίησα τα δύο μου λεπτά. Πρόεδρος, χρησιμοποιήσατε ένα λεπτό και 15 δευτερόλεπτα για να είμαστε ε, ακριβείς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα είμαι πολύ σύντομος. Ε, αυτή είναι η έκθεση για τις δικές μας δραστηριότητες ε, με βάση τον κανονισμό που υπάρχει στο Κοινοβούλιο. Οι δικές μου οι ε, παρατηρήσεις είναι περισσότερο οι φιλικές παρατηρήσεις ενός παρατηρητή. Φιλικές ε, γιατί δουλεύω βασικά για σας και όλα αυτά είναι πολύ καλά για σας και για μένα. Εντυπωσιάστηκα από αυτά που είπε ο κύριος Μίτσελ. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό που έθιξε ο κύριος Μίτσελ και αυτό το έχουμε συζητήσει και εμείς με συναδέλφους της Κομισιόν πολλές περιπτώσεις. Πολύ σημαντικό αυτό που είπε. Το δεύτερο και τελευταίο που θέλω να πω είναι ότι ήδη με την περσινή έκθεση από τον κύριο Μπουσετήλ οι τροπολογίες του κυρίου Μπουσετήλ πιο συγκεκριμένα ε, προσπάθησαν να δώσουν έτσι μια συγκεκριμένη μορφή στις δραστηριότητες σας. Φαντάζομαι ενστικτοδός θα γνωρίζετε τι είναι το ε, καλύτερο που οφείλετε να κάνετε. Ε, όμως ε, είναι καλό να βλέπει κανείς ε, ξεκάθαρα ε, ποιες είναι οι δραστηριότητες που απέδωσαν αξία στην Επιτροπή και νομίζω αυτή η έκθεση συμβάλλει προς το να ακολουθεί περισσότερο αυτή η κατεύθυνση και είναι καλό αυτό και ο διαμεσολαβητής το ίδιο κάνει και με τη δική του την ετήσια έκθεση βλέπουμε ότι τα καταφέρνει πολύ καλά στο να αποκτήσει περισσότερους πόρους για τις δραστηριότητες του και αυτή η έκθεση ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση και πολύ σωστά κάνει. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ε, η κυρία Μακκίνες, ε, ευχαριστώ όλους τους ε, συναδέλφους για τα σχόλιά τους και την Επιτροπή και επιτρέψτε με πολύ σύντομα να τοποθετηθώ. Νομίζω ότι στο θέμα της Equitable Life θα πρέπει να προσθεθεί κάποια παράγραφος. Ε, θα περιμένω ότι θα πει ο πρόεδρος στο Κοινοβούλιο. Ε, όσον αφορά το εκεί θα προσθέσουμε και κάποια γεωγραφικής φύσεως θέματα θα το αλλάξουμε λιγάκι εξάλλου πολύ σημαντικό αυτό που είπατε ότι είναι πολύ δύσκολο να υπάρχει αστυνόμευση εμείς ε, θέλουμε να δούμε τη δυνατότητα ε, στους ε, αναφέροντας ότι υπάρχει το στοιχείο της ε, αμφιβολίας. Όσον αφορά την Επιτροπή για την Equitable Life, ε, όλοι όσοι ήρθαν στην Επιτροπή ξέρουν ότι δεν μπορούμε να δώσουμε χρήματα στους ενδιαφερόμενους αλλά να τους παρουσιάσουμε μια δίκαιη έκθεση. Όσον αφορά τα σχόλια του κυρίου Μαυρομάτη για τα κράτη-μέλη βεβαίως και αυτά θα τα λάβουμε υπόψη μας και για τα θέματα που είπε ο Σερ Ρόμπερτς για το προσωπικό ε, πράγματι αυτά ε, θα ληφθούν υπόψη. Εγώ θα χαρώ ε, να κατεθούν τροπολογίες στην έκθεση ε, και ίσως μπορείτε να μου πείτε, να μου το υπενθυμίσετε πότε θα υπάρξει και η σχετική ψηφοφορία Ίσως μπορεί αυτό να το κάνει η γραμματεία. Κοιτάξτε, στις 12 Μαρτίου, στις 12 το μεσημέρι θα είναι η ψηφοφορία και μέχρι τότε ε, μπορούν, μάλλον, μέχρι τότε μπορούν να κατευθύνουν τροπολογίες και στις 31 Μαρτίου είναι η ψηφοφορία. Και εγώ θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ και να επισημάνω κάτι που είπε ο κ. Φλόιντ. Είπατε ότι θα είναι πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε ε, κάποια στατιστικά δεδομένα για τη συνέπεια. Αυτό είναι πολύ δύσκολο η εμπειρία μου των τελευταίων πέντε ετών έδειξε ότι ε, δεν μπορούμε ε, αμέσως να βρούμε τη λύση. Μπορούμε να την προβάλλουμε ως προοπτική αν θέλετε, αλλά το να υπάρχει έτσι κάποια συστηματική παρακολούθηση και έχουμε πρόβλημα. Πριν από τέσσερα χρόνια ασχοληθήκαμε με τη διακριτική μεταχείριση ε, των ε, επιχειρήσεων των νέων κρατών μελών που δραστηριοποιήθηκαν στα παλαιά κράτη-μέλη. Εκεί κατατέθηκε μία ολόκληρη σειρά αναφορών. Εμείς ενημερώσαμε τις αρμόδιες υπηρεσίες και πρέπει να σας πω ότι δεν κατατέθηκαν άλλες ε, σχετικές αναφορές. Αυτό λοιπόν μας οδηγεί στο να ελπίζουμε ότι εμείς δραστηριοποιηθήκαμε και αυτό έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ε, πάνω από τέσσερα χρόνια ασχολούμεθα με τα γερμανικά κέντρα νεότητας ε, και υπάρχουν ε, κάποιες ενδείξεις από τους δικηγόρους και από τους γονείς ότι βελτιώθηκε η κατάσταση. Όταν λοιπόν κάποιος ε, έρχεται σε εμά ε, και καταθέτει μία αναφορά ή κάνει μία καταγγελία για μία συγκεκριμένη υπόθεση, τότε αυτό δεν σημαίνει ότι διεκπεραιώνεται το όλο θέμα, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ε, η τάση ε, που προκύπτει είναι ότι κάτι γίνεται. Και το γεγονός ότι προέκυψε μια βελτίωση με τα κέντρα νεότητας, νομίζω αυτό είναι ικανοποιητικό. Κατά πόσον τώρα μπορούμε να έχουμε στατιστικά δεδομένα για να τεκμηριώσουμε αυτή την άποψή μας, εδώ πρέπει να πω αυτό με ξεπερνάει. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι διαπιστώνουμε μια τάση. Η κυρία Μακίνες αναφέρθηκε στην έκθεση για τον αγωγό North Stream. Σουηδική κυβέρνηση επικαλείται συνεχώς ε, στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ε, έκθεσή μας. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα κατασκευαστεί ο αγωγός ή όχι. Εκείνο που γνωρίζουμε όμως είναι ότι η δική μας η έκθεση τελικά κατέστη εργαλείο στα χέρια εκείνων οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτήν την ε, επένδυση επιφυλακτικά. Άρα δηλαδή καταλαβαίνετε καταλήγω στο ότι μία παρακολούθηση των εξελίξεων, ε, των δραστηριοτήτων μας ε, για πολλά χρόνια μας οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα. Πάμε στην επόμενη αναφορά που αφορά την κυρία Αναστασία Γάκη, η οποία η κυρία Γάκη είναι παρούσα και έχετε παρακαλώ πέντε λεπτά στη διάθεσή σας. Ναι, ε, αγαπητές μου κυρίες και κύριοι, κατα... αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Καταρχήν σας ευχαριστώ που βρίσκομαι εδώ. Ε, θα μπω κατευθείαν στον θέμα. Θα γνωρίζετε όλοι σας σίγουρα το άρθρο 6.1 ε, και 2 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το οποίο τέθηκε σε ισχύ στην χώρα μου, στην Ελλάδα, με το νομοθετικό διάταμο του 78, μάλιστα με στεγματική ισχύ. Επίσης υπάρχει ο κανονισμός 1348 του 2000 που κυρώθηκε στην Ελλάδα από τις 31 Τρίτου του 2003 που αφορά τις επιδόσεις για ποινικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όλα αυτά δεν ξέρω για ποιο λόγο. Η κυρία 18η ανακρίτρια Αθηνών, κυρία Ιωάννα Στρατσιάνη, την περίοδο του Μαρτίου του 2006 δεν τα έλαβε καθόλου υπόψη της. Ε, υπήρχε ο μηνυτής, κατά του πατέρα μου τον οποίον εκπροσωπώ, παρόλο που στις 28 Τρίτου του 2006 της εγχείρησε ένα ακριβώς σχεδιάγραμμα της κατοικίας μου στον Τίστελοφ, Παρόλο που υπήρχαν ε, οι καταθέσεις του από τις 13 του 2006 και από τις 14 Τρίτου του 2006, όπως και τις κόρες του μάρτυρα, από όπου αποδεικνυόταν πολύ καλά η κατοικία μας στο Σοντίστελντοφ, παρόλα αυτά η 18η ανακρίτρια στέρνει κλήσει σε διευθύνσεις που ποτέ έμεινε ο πατέρας μου, με εντολή να θυροκολούνται είτε σε ένα κλειστό σπίτι ή να επιστρέφουν πίσω όσο του διαμονής, και είχε ω συνέπεια να βγουν εντάλματα συλλήψεως ει βάρος του πατέρα μου και όταν πήγε να παραλάβει η ταυτότητά του συλλαμβάνεται, δεν μαθαίνει το λόγο τη σύλληψή του παρά μόνο μετά από πέντε μέρες και οδηγείται σε δύο μήνες σε μία δίκη και καταδικάζεται ε, για 12 ε, χρόνια. Δεν θα πω στο ουσιαστικό ε, θέμα της δίκης που δεν υπήρχε ούτε μία έστω ένδειξη ενοχής εις βάρος του Επικεντρώνομαι περισσότερο στην τυπική διαδικασία που δεν τηρήθηκε και θα ήθελα εδώ πέρα να κάνω μια πολύ μικρή παρένθεση. Ε, όλη η δικογραφία την παρουσίασε ένας φίλος μας στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, συγκεκριμένα στις 28 Ενδεκάτου του 2008. Διαβάστηκε η δικογραφία, ο κύριος Υπουργός Δικαιοσύνης ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά μου, Ήθελα να μάθει τα ονόματα δικαστιών που γινόταν στην αίτηση αναστολής ποινή του πατέρα μου για τι 15 Δεκάτου, για να τον βγάλουν έξω να μην τυραννείται τελικά ένας αθώος μέσα στη φυλακή και στις 15 η ώρα 3 το μεσημέρι ο πρόεδρος Πρωτεδικών Αθηνών τηλεφωνεί τον κύριο Γενικό Γραμματέα Αναγνωστόπουλο του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του λέει «Δεν θα αφήσετε έξω το γάκι τηλέμαχο, η υπόθεση είναι δικά μας, μην ανακατεύεστε στα ξένα χωράφια, γιατί θα καούν τα χέρια σας». Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Επιθυμώ, γιατί με τον Υπουργό Δικαιοσύνη δεν μπορώ να έχω καμία συνομιλία. Του έχω στείλει επανειλημμένε αναφορέ, δεν μου έχει απαντήσει. Όπω ο κύριο Αγγελέα του Αρίου Πάγου, κύριο Ανιδά. Και ειλικρινά λυπάμαι που έχω φτάσει εδώ για να φέρω αυτό το πρόβλημα. Τι επιθυμώ από εσά. Ε, το δικαστήριο του πατέρα μου του αφετίου, που ουσιαστικά και το πρώτο βαθμού δεν έχει καμία κανένα νόμια, βρίσκεται στη, θα γίνει στις 20 Δευτέρου του 2009, τώρα σε 10 μέρες. Επειδή δεν πιστεύουμε την ελληνική δικαιοσύνη και με όλα αυτά που έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν την εμπιστεύομαι, θα ήθελα, εάν είναι εφικτό ένας εκπρόσωπος, να παραστεί στη δίκη. Διότι πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχιστεί αυτό σε εσβάρος ενός αθώου 74 χρονών ανθρώπου και κανείς μα κανείς δεν συγκινείται. Υπάρχει μια πληροφορία ότι του μηνυτή ο Πατζανάκης είναι γενικός διευθυντής του κυρίου Κόκαλη, ο οποίος έχει προσωπικές σχέσεις με πολλούς δικαστέ στην Ελλάδα. Αυτά που σταλώ προφορικά μπορώ να σα τα πω και γραπτά και να τα υπογράψω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορείτε να ακούσετε τον συνάδελφό μου κύριο Ανδρέο Χάινε θα ήθελα να συμπληρώσω τα εξή από νομική πλευρά. Ε, νόημα αυτής της ρύθμισης για τις επιδόσεις των Ελλήνων που διαμένουν στο εξωτερικό, οι οποίοι μέσω αυτής της διάταξης εξισώνονται με όσους μένουν με, με τους είναι σαφές ότι ένας Έλληνας ο οποίος διαμένει στο Ντούσελντορφ εδώ και 14 χρόνια όταν ξεκινάει μια διαδικασία εναντίον του θα πρέπει να γίνεται η επίδοση αυτού του εγγράφου στη Γερμανία. Γιατί αυτό έχει το νόημα πρώτον να ενημερώνεται εγκαίρως ο ενδιαφερόμενος και να μπορέσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων υπεράσπισής του. Και, στο μετρο... και ο κύριος Γάγκης λόγω αυτού του... αυτής της παράληψης για την οποία δεν υπάρχει απολύτως καμία εξήγηση γιατί ήταν γνωστό ότι ο κ. Γάκης ε, διαμένει στη Γερμανία και οι αστυνομικές ε, αρχές ε, παρακλήθησαν να βρουν τη διεύθυνση του κυρίου Γάκη. Ήταν αποδειγμένο λοιπόν ότι διαμένει ο κύριος Γάκης στη Γερμανία. Δεν μπορούμε λοιπόν να κατανοήσουμε το πώς η ανακρίτρια λίγες μέρες μετά εξέδωσε ένα ένταλμα σύλληψης του κυρίου Γάκη το οποίο τελικά έγινε εκτελεστό λίγες μέρες μετά. Και μπορώ να καταλάβω τις ανησυχίες της οικογένειας που, γιατί ο, ο πατέρας αυτός ε, βρίσκεται, κρατείται εδώ και 18 μήνες, είναι αρκετά μεγαλη ηλικία, η κατάσταση υγείας σου δεν είναι καλή και υπάρχουν πολλές ανησυχίες εκ μέρους της οικογένειας ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει για πολύ καιρό εάν παραμείνει ακόμα στη φυλακή. Ευχαριστώ. Ο κ. Τόμας από την Κομισιόν. Ε, ε, European Commission... Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καμία εξουσία να παρέμβει στην ε, καθημερινή διαχείριση του δικαστικού συστήματος ή ουδήποτε κράτους μέλους. Οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρέουν από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 33 της συνθήκης αυτής προβλέπει ότι τα κράτη-μέλη τα ίδια είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση της τάξης και του νόμου στην επικράτειά τους. Επομένως, το θέμα αυτό είναι αποκλειστικής ελληνικής αρμοδιότητας και η Κομισιόν δεν έχει τίποτα να προσθέσει. Ευχαριστώ. Ε, Τώρα, pan Κύριος Γεωργίου και μετά κυρία μου θα σας το λόγο. Κυρία Γάκη. Πρόεδρε, επειδή βρισκόμεθα ενώπιον προφανούς περιπτώσεως μη συμμορφώσεως των ελληνικών αρχών με τον κανονισμό 1348 του 2000 όπως ανεφέρθηκε όλα του Συμβουλίου περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως στα κράτη-μέλη δικαστικών και εξωδικών πράξεων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη του άρθρου 33 και 35 παράγραφος 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή κύριε Πρόεδρε νόμιμος δίκη προϋποθέτει και απαιτεί νόμιμον επίδοση νομίμου κλητεύσεως θεωρώ ότι θα είναι αναγκαίων ηθικών και δίκαιων ε, να επανεξετάσουμε το φάκελο ΓΑΤΚΙ, δεδομένου ότι η αρμοδία χειρίστρια παρά το γεγονός ότι το γνώστης της διευθύνσεως του αναφερομένου ο οποίος από δεκαετίες ή από τη δεκαετία του 60 ε, διαμένει μονίμωση στο εξωτερικό συμφώνως προς έγγραφον βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής η ανακρίτρια επέλεξε να τυχοκολλήσει την ειδοποίηση σε διεύθυνση η την οποία ο μηνιόμενος και η οικογένειά του ουδέποτε χρησιμοποίησε. Δεν έμεινε ποτέ εκεί. Επειδή δεν δίναμε να φανταστώ ότι βρισκόμεθα προδολίου ενεργεία, αυτό δεν το δέχομαι, παρακαλώ να εξεταστεί από την Επιτροπή μα, το ενδεχόμενο σοβαρού ανθρωπίνου σφάλματο. Ε, και βεβαίω η Κομισιόν θεωρεί ότι η αναφορά εμπίπτει στι αποκλειστικέ αρμοδιότητε των ελληνικών αρχών. Αλλά βεβαίω ο παραπονούμενο πολίτη εμπίπτει στην αρμοδιότητα τη λογική και της βασικής αρχής της απονομής της δικαιοσύνης η οποία απαιτεί προετοιμασία και νόμιμον κλήτευση του ενδιαφερομένου προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της απονομής του δικαίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Proszę Państwa, Πρόεδρος, πρόκειται για μια διάρρουσα κατάσταση θα έλεγα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Κομισιόν έχει αρμοδιότητα για δικαστικά θέματα. Όμως, από αυτά που είπατε για την έλλειψη κοινοποίησης και από αυτά που είπε και ο κύριος Γεωργίου προκύπτει ότι χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις για το θέμα αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι θα μπορούσαμε να γράψουμε και να ζητήσουμε αυτές τις διευκρινήσεις και ελπίζουμε ότι θα εξομαλυνθούν τα πράγματα. Θέλετε το λόγο, σύντομα παρακαλώ. Τον έχετε. Έχετε το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα με έχει καλύψει ο κύριος ε, Γεωργίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Υπάρχει ένας κανονισμός της Κομισιόν. Έχουμε τώρα αυτή την ενημέρωση ότι υπάρχει σχετικό κανονισμός. Δηλαδή υπάρχουν διάβλοι ακόμα για την ε, Επιτροπή. Έχουμε ενημέρωση στο φάκελό μας για αυτόν τον κανονισμό 1348 του 2000. Κομισιόν, πώς θέλετε να αναφέρετε τίποτα για αυτόν τον κανονισμό. Όχι, Πρόεδρε. Θεωρώ ότι το θέμα είναι αμυγός ελληνικό. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα περαιτέρω. Πρόεδρος. Πολύ ωραία, θα κάνουμε αυτό που σας είπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους αναφέροντες. Περνάμε τώρα. Παρακαλώ. Λέξη ε. μόνο κύριε Πρόεδρε, αναφερόμενος στον κύριο της Κομισιόν. Ε, βεβαίως ναι. μιλήσαμε για το ενδεχόμενο ανθρωπίνου λάθους. Βεβαίως αποκλείσαμε την περίπτωση δόλου. Αλλά εάν έτσι ξηρά κλείνουμε ένα φάκελο και λέμε ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι οι ελληνικές αρχές έχουν την απόλυτη αρμοδιότητα, τότε δεν αντιλαμβάνουμε την παρουσία τη δική μας εδώ ως επιτροπή. Przepraszam Συγγνώμη, αλλά δεν κλείσαμε αυτή την αναφορά. Η αναφορά παραμένει ανοιχτή. Α δώσουμε το λόγο στην εκπρόσωπο τη Ελληνική Μόνιμη αντιπροσωπείας. Κύριε Πρόεδρε, ε, επειδή προφανώς δεν γνωρίζετε, είμαι από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία. Ε, είμαι δικαστής αποσπασμένη στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στα θέματα του, της, αστικής συνεργασίας, της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις. Ο κανονισμός στον οποίο αναφερόμαστε είναι ένας κανονισμός ο οποίος, όπως λέει και ο τίτλος του, αφορά επίδοση σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Εάν δείτε το σχετικό άρθρο του πεδίου εφαρμογής αποκλείονται διοικητικές και ποινικέ υποθέσεις. Επομένως, η ανακρίτρια δεν μπορούσε να κάνει επίδοση με χρήση του κανονισμού αυτού. Απαγορεύεται. Από εκεί και πέρα, εάν θα έπρεπε να κάνει επίδοση με βάση διεθνείς συμβάσεις με τις οποίες γίνεται η κοινοποίηση στο εσωτερικό, αυτό φαντάζομαι ότι το ήλεγξε. Φαντάζομαι ότι αν η ίδια ήταν εδώ θα μπορούσε να μας δώσει και περισσότερες πληροφορίες για το πώς δούλεψε την υπόθεση. Ναι, κατακλείδη μόνο να σας πω ότι τα δικαστήρια είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο θέμα της εμφάνισης και της κλήσης του κατηγορουμένου. Ο δε κατηγορούμενος ή οποιοδήποτε πολίτης γνωρίζει ότι υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί για κάτι, μπορεί και αυτόκλητα μόνος του, χωρίς κλίση, να εμφανιστεί και να πει την άποψή του. Από ό,τι κατάλαβα η κυρία Γάκη έδωσε, είπε τη διεύθυνσή της. Άρα γνώριζε ότι για κάποιο λόγο ζητούσαν τον πατέρα της. Ο πατέρας της και αυτόκλητα μόνος του μπορούσε να παρουσιαστεί. Βέβαια δεν επεμβαίνω στην ουσία της υπόθεσης, αλλά γι' αυτό ακριβώς το λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι είναι θέμα εσωτερικής ε, ελληνικής νομοθεσίας. Ευχαριστώ. Tak, więc proszę Pani wspomniała, że gdyby sędzia była tutaj, to by mogła to wszystko wyjaśnić. My nie oczekujemy, że sędzia przyjdzie. Πρόεδρος. Είπατε ότι ένας δικαστής θα μπορούσε να μας εξηγήσει όλα αυτά. Αλλά αυτό δεν είναι... Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε μάλλον είναι να γράψουμε σε ένα δικαστή, να μας απαντήσει και να έχουμε όλες τις εξηγήσεις. Πάμε τώρα στο σημείο 16, αναφορά 440 το 2006. Η Ελίζα Πεθγκαρουφάλου έχει το λόγο. Καλημέρα. Αυτή η αναφορά αφορά την ε, δυνατότητα που έχει παραχώρησης ε, κρατικών ενισχύσεων από το Μαλτέζικο κράτος με προδημισιακές τιμές. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχει τέτοιο ενδιαφέρον από τους stakeholders, επιτρέψουμε αυτή την αγγλική έκφραση, ούτω ώστε οι κανόνες κανονισμού να εφαρμόζονται σωστά. Επίσης, η κατάσταση με βάση τα όσα λέει αναφορά τροποποιήθηκε. Γιατί από ό,τι βλέπουμε τον Οκτώβριο του 2008 αναθεωρήθηκε τελείως το σύστημα των τιμολογίων στη Μάλτα αυτή η υπερβολική τιμή για, το, για το πετρέλαιο πλέον δεν υφίσταται. Παρακαλώ να μιλάτε στους διαδρόμους. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Γιατί δεν έχουμε τέτοια στοιχεία που να πιστοποιούν κάτι τέτοιο, ότι υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Θα πρότεινα στους αναφέροντες να μας δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία, ε, γιατί όπως σας είπα έχουν αλλάξει και τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη κατάσταση, η Κομισιόν είχε ήδη εκφραστεί. Είχαμε πει ότι δεν είχαμε αρκετούς, αρκετά στοιχεία για να αποφανθούμε ότι πρόκειται για κρατικές ενισχύσεις. Από την άλλη, ο καλύτερος τρόπος για να κυρώσουμε οποιασδήποτε παραβάσει ό,τι αφορά τις ε, κρατικές ενισχύσεις δεν είναι η οδός των αναφορών. Αν και βέβαια οι αναφορές ουσιαστικά ε, συνιστούν μια πολιτική διαφήμιση και είναι χρήσιμο κάτι τέτοιο σε περίπτωση που υπάρχουν παραβιάσεις. Έχουμε όμως διαδικασίες οι οποίες είναι πολύ πιο συγκεκριμένες για τις κρατικές ενισχύσεις και που πρέπει να ακολουθηθούν. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαμε να παραπέμψουμε επί παραβάση ένα κράτος μέλος, το οποίο είναι αναγκασμένο να μας δώσει όλα τα στοιχεία για να μας πείσει πώς, έχει, πώς έχουν τα πράγματα. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερα στοιχεία και θα θέλαμε ενδεχομένω να γίνει μια καταγγελία ότι υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις στη Μάλτα και θα πρέπει κυρίως να σταθούμε σε κάποιες ουσιαστικέ ερωτήσεις για μας. Δηλαδή θέλουμε να καταλάβουμε τι αντικειμενικά στοιχεία υπάρχουν που να μας πείθουν ότι όντως υπάρχουν κρατικές ενισχύσεις. Γιατί συχνά υπάρχουν λόγοι που δικαιολογούν ε, διαφορετικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά αντικειμενικοί λόγοι. Πολύ ωραία. Κομισιόν, μπορούμε να κλείσουμε αυτή την αναφορά λοιπόν. Πάμε στο σημείο 17. Αναφορά 951 του 2004 η κυρία Μόνικα Βαλόρτσικ. Η δική μας η αναφορά αφορά στο άρθρο ε, που έχει σχέση με το ΦΠΑ, το άρθρο 77. Εδώ λοιπόν η ε, Κομισιόν θα το πω αλλιώς. Το 2008 ε, στάλει μία αναφορά για να λυθεί το θέμα του ΦΠΑ. Δόθηκε μία απάντηση από, τον από την Πολωνία και από εκεί απορρέει ότι προετοιμάζονται νέες διατάξεις. Τον Ιούλιο του 2008 το Ευρωπαϊκό ε, δικαστήριο ε, αποφάνθηκε στην περίπτωση της Αλήσιας Οσνόσκα και το δικαστήριο καταλήγει στο ότι η ε, παράταση καταβολής του ΦΠΑ σε 180 ημέρες δεν σημαίνει ότι συνεπάγεται και την καταβολή εγγύηση σε ύψους 250.000 ζλότη. Αυτό είναι αντισυνταγματικό. Κατόπιν λοιπόν η πολωνική κυβέρνηση έστειλε μια επιστολή ερωτώντας τι είδους ε, μέτρα θα πρέπει ληφθούν για να προσαρμοστεί ε, το πολωνικό δίκαιο ΦΠΑ στο ε, κοινοτικό δίκαιο. Αργότερα λάβαμε μία απάντηση με την ανακοίνωση ότι το Νοέμβριο του 2008 οι διατάξεις του άρθρου 57 που ρυθμίζουν αυτό το θέμα. Οι διατάξεις αυτές ε, καταργήθηκαν από το, ε, την νομοθετική διάταξη της Πολωνίας ε, περί ΦΠΑ. Και προσαρμογή της διάταξης τέθησε σε ισχύ έτσι ώστε να λυθεί το θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να σας ρωτήσω το εξής. Όλα αυτά σημαίνουν ότι τώρα πλέον δεν κρίνεται απαραίτητο να καταβάλλεται αυτή η εγγύηση, αυτό το αστρονομικό ποσό ή τι γίνεται, επιστρέφεται, φυπία, τι ακριβώς κάνετε, δεν καταβάλλει την εγγύηση, πώς ακριβώς έχει η τι γινεται επιστρεφεται ΦΠΑ. τι ακριβως κανετε δεν καταβαλλει την εγγυηση πως ακριβως εχει η κατασταση Και θα ήθελα Επίσης να σας ε, παρακαλέσω να μας στείλετε μια επιστολή ενδεχομένως αύριο γιατί για μας το όλο θέμα είναι πολύ σημαντικό. Ε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που επιληφθήκατε αυτού του θέματος γιατί για πάρα πολλές πολωνικές επιχειρήσεις ε, είναι θέμα αρχής. Το όλο θέμα διαρκεί εδώ και τέσσερα χρόνια και πρέπει να σας πω ότι το παλεύουμε εδώ και πολύ καιρό. Απευθυνθήκαμε στις πολωνικές αρχές, ε, στους αναφέροντες. Πραγματικά θα σας ήμουν ευγνώμων εάν ήδη αύριο μπορούσατε να μας στείλετε μία επίσημη επιστολή που θα περιλαμβάνει όλες αυτές τις πληροφορίες. Γιατί οι πληροφορίες που μας δόθησαν ε, σε γραπτή μορφή είναι πλέον παροχημένες κύριε Πρόεδρε. Θα ακούτε ε, μάλλον ότι είμαι κρυωμένη και δεν θα προλάβω μέχρι αύριο. Μπορώ μέχρι τέλος εβδομάδας. Εντάξει, μέχρι τέλος εβδομάδας μπορείτε να στείλετε την επιστολή αυτή στη γραμματεία. Άρα δεν κλείνει το θέμα τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η αναφορά ε, παραμένει ανοιχτή. Βλέπω ότι τα μέλη της ε, Επιτροπής ε, που βρίσκονται στην αίθουσα συμφωνούν και ως εκ τούτου μου επιτρέπεται να διακόψω τη συνεδρίαση μέχρι αύριο το πρωί στις 9 όπου θα συνεδριάσουν οι συντονιστές και στις 10 θα ξεκινήσει η κανονική συνεδρίαση. Σας ευχαριστούμε πολύ.